Colleagues, good afternoon. Can I bring the... Πάμε αγαπητοί συνάδελφοι, καλό απόγευμα. Αρχίζει η συνεδρία της Επιτροπής Μεταφορών αλλά και Τουρισμού. Έχετε την ημερήσια διάταξη, το σχέδιο τη τουλάχιστον. Is that any noisier, Jackie? No? Okay. Okay, can I the adoption of the draft agenda is... Έγκριση ημερήσια διάταξη, είστε ικανοποιημένοι από τη ημερήσια διάταξη. Ωραία. Περνάμε στην έγκριση των πρακτικών τη 28η Φεβρουαρίου και τη 14η με 16η Μαρτίου του Ενιστότο. Και αυτά σα αρέσουν, εντάξει, είσαστε ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ ανακοίνωση της νέας θέσης του Συμβουλίου σε σχέση με τον κανόνα ε, το άρθρο 63 του κανονισμού και μετά από την ανακοίνωση της θέσης του Συμβουλίου στην Ολομέλεια στις 24 Μαρτίου 2011 για την διαμεθοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για την ασφάλεια, οδική ασφάλεια σε ό,τι αφορά διαμεθοριακή, διαμεθοριακά δικήματα με εισηγήτρια την κυρία Αιάλα Σέντερ, το Συμβούλιο θα, η θέση του Συμβουλίου θα παρουσιαστεί ως πρώτο σημείο στην ημέρησια διάταξη. Η έκθεση της κυρίας Αγιάλα Σέντερ θα συζητηθεί αύριο το απόγευμα στις 3 ώρα, αλλά όλα αυτά πρέπει να σας τα ανακοινώσω σήμερα. Το επόμενο σημείο, εξέταση τροπολογιών για την επιβολή τελών σε βαρέα φορτικά για τη χρήση ορισμένων υποδομών, η λεγόμενη Ευρωβινιέτα. Ο κύριος Αλχαντράουι είναι εισηγητής και έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα αγαπητοί συνάδελφοι να ευχαριστήσω καταρχήν όλους αυτούς οι οποίοι τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθούσαν με μεγάλο ενδιαφέρον τα θέματα αυτά και συζήτησαν μαζί μου για να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες και να μπορέσουμε να συγκεράσουμε τις απόψεις μας ώστε να έχουμε μια ενιαία θέση εναντί του Συμβουλίου. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους σκιώδεις εισηγητές, οι οποίοι έκαναν μεγάλη προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Γνωρίζω απόλυτα το ότι κανείς δεν μπορεί να είναι 100% ικανοποιημένος με αυτή την συμβαστική θέση. Ορισμένοι θεωρούν ότι είναι υπερβολικά φιλόδοξη, άλλοι όχι αρκετά φιλόδοξη. Και είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε από το Συμβούλιο δεδομένων των δυσκολιών και δεδομένων των διαφορών απόψεων μέσα στο Συμβούλιο. Ξέρουμε ότι ήταν η συχνότατη πλειοψηφία με την οποία ενεκρίθη η κοινή θέση του Συμβουλίου. Υπάρχει πόλωση για πέντε ζητήματα. Το ένα είναι το θέμα του εξωτερικού κόστους, εμείς θεωρούμε ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να συνδέεται το θέμα αυτό με μεγαλύτερη ευκαμψία σε ό,τι αφορά τη φορολογία για τις υποδομές. Έλα ρε Μισλιν, μίλα κανονικά. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ουδετερότητα σε επίπεδο προϋπολογισμού για τα μέτρα αυτά και νομίζω ότι και σε αυτό το σημείο υπήρξε μια συμφωνία. Το δεύτερο θέμα το οποίο ήταν επίμαχο ήταν το θέμα της εμβέλειας αυτής της, αυτού του νομοθετήματος, διότι η άποψή μας ήταν ότι όταν αφορά το το βάρος των φορτηγών, θα πρέπει να καλύπτει όλα τα φορτηγά από 3,5 τόνους και άνω. Αυτό είναι όμως δύσκολο σε ορισμένα κράτη-μέλη που θέλουν να διατηρήσουν τις ιστορικές τωρινές ε, ρυθμίσεις και να ξεκινήσουν αργότερα με την επιβολή ενιαίων ρυθμίσεων. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε τίποτα εδώ. Χρειάζεται πραγματισμός και χρειάζεται και μια σωστή επιλογή διατύπωσης. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε ότι το όριο των 3,5 τόνων θα πρέπει να ισχύσει εν καιρό, αλλά μπορούμε να το εξετάσουμε περαιτέρω το θέμα αυτό με το Συμβούλιο. Το τρίτο σημείο είναι το θέμα των ε, οχημάτων Euro 6 για τα οποία θα ισχύσει σε ορισμένε περιπτώσει σε τρία χρόνια, σε άλλε σε τέσσερα χρόνια. Άλλε άλλες κατηγορίε αυτοκινήτων θα έχουν χρόνο μετάβαση δύο χρόνων μονάχα. Και επίσης το θέμα των, ε, ε, της καταλογισμού εξωτερικού κόστους για δημιουργία σειράγκων στα βουνά, για διαβάσεις κτλ. Όλα αυτά έχουν αναφερθεί ήδη με το Συμβούλιο. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τα αυτοκίνητα κατηγορίας Euro 1, 2, 3 και 4 και πιστεύω ότι εδώ μπορούμε να επιλέξουμε μία ενδιάμεση ε, κατάσταση ώστε να για τα 1, 2 και 3. Ευρώ 1, 2 και 3. Το επόμενο θέμα είναι τα επόμενα βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν. Και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το λεγόμενο earmarking. Ο προσδιορισμός των εσόδων για συγκεκριμένους στόχους. Το Συμβούλιο εδώ ήθελε απλώς να υπάρχει μια σύσταση προς την κατεύθυνση του προσδιορισμού, ενώ το Κοινοβούλιο θα ήθελε τα έσοδα τα οποία προέρχονται από τα τέλη των φορτηγών να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία μεταφορικών υποδομών. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο σε επίπεδο πρώτης ανάγνωσης να τονίσουμε την θέση μας για τον προσδιορισμό όλων αυτών των εσόδων, των τελών. Αυτή είναι φυσικά μια αρχική διαπραγματική, διαπραγματευτική θέση και ίσως θα καταλήξουμε και σε μια συμβιβαστική λύση και πολλοί συνάδελφοι έχουν καταθέσει τροπολογίες οι οποίες προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια καλύτερη προσέγγιση προς τη θέση του Συμβουλίου και ακολουθείται από ορισμένους η διατύπωση της οδηγίας ΕΤΕΕΣ. Ίσως λοιπόν μπορούμε να κατευθυνθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Εγώ όμως προτείνω να μην το πράξουμε αυτό ακόμα να παραμείνουμε πιστοί σε μια θέση απόλυτου και υποχρεωτικού προσδιορισμού, τουλάχιστον προς το παρόν. Αυτά λοιπόν για τους σκιώδεις και ε, τους συναδέλφους. Με τους σκιώδεις εισηγητές έχουμε διεξέλθει όλες τις τροπολογίες. και έχουμε ζητήσει από την Κομισιόν να υπάρξει και ένα εγκόλπιο το οποίο θα δίδεται στους οδηγούς ώστε οι χρήστες να καταλαβαίνουν τι προκύπτει από αυτή την οδηγία, πώς θα πρέπει να εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες και ο στόχος μας επίσης με τις τροπολογίες μας ήταν να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη σαφήνεια και πολλοί συνάδελφοι Θέλησα να τονίσουν την ε, διαλειτουργικότητα των διαφόρων μορφών μεταφοράς. Εδώ κατατέθηκα λοιπόν τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν και τροπολογίες επίσης, για τις οποίες εγώ έχω κρατήσει μια αρνητική στάση. Είναι τροπολογίες που μου φαίνονται ότι είναι περιτές, ή αποκλίνουν πολύ από την συμβιβαστική θέση την οποία έχουμε προσπαθήσει να συμπήξουμε. Και προχωρούν προς την κατεύθυνση της ε, πλήρους εσωτερικοποίησης του κόστους ή πάνε προς την κατεύθυνση της μη εσωτερικοποίησης του κόστους, δηλαδή πηγαίνουν προς τα άκρα. Αυτή είναι λοιπόν η η διαφαινόμενη συμφωνία αυτή τη στιγμή για το θέμα αυτό, το οποίο είναι ένα πολύπλοκο θέμα, το οποίο είναι πολιτικά ευαίσθητο. Πιστεύω λοιπόν ότι με το πακέτο αυτό το οποίο έχουμε ενώπιόν μας έχουμε επιτύχει μια πολύ καλή βάση για να βελτιώσουμε την κοινή θέση του Συμβουλίου και να καταλήξουμε σε μια λύση πριν από το καλοκαίρι. Και στη συνέχεια τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να εξετάσουμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτού του νομοθετήματος και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε ενώπιον μας τώρα είναι το ελάχιστο. Για πρώτη φορά εξασφαλίστε ότι το εξωτερικό κόστος εν μέρη τουλάχιστον θα εσωτερικοποιείται. Αυτά ήθελα να πω λοιπόν και θα ήθελα να ακούσω και τις απόψεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βορτμαν, Κούλ, εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, Ρίχνοντα μια ματιά στι ε, τροπολογίε. Πιστεύω θα διαπιστώσατε, και δεδομένου και ποιος έχει καταθέσει, ότι έγινε μια μάλλον έντονη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για τις ε, προτάσει που θα καταθέταμε στις διαπραγματεύσεις μας με το Συμβούλιο. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί στάθηκε σε ορισμένα κέρια σημεία, κέρια για μας σημεία και δέχθηκε ε, να προχωρήσει σε συμβασμό μαζί μας έτσι ώστε να μπορέσουμε και στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο να επιμείνουμε στις δικές μας προτεραιότητες, τις προτεραιότητες που θεωρεί η ομάδα μας ως τις πιο σημαντικές με την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πρόοδο στα δικά μας θέματα. Έτσι λοιπόν, διαλειτουργικότητα. Ε, συστήματα διοδίων που έχουν εισαγάγει τα περισσότερα πλέον κράτη-μέλη και τα υπόλοιπα ακόμη συνεχίζουν από ό,τι φαίνεται. Ευτυχώς η διαλειτουργικότητα λοιπόν δεν μένει στα χαρτιά, προχωρεί στην ουσία και θεωρώ ότι είναι πολύ καλό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο εμένει στα πράγματα αυτά. Επίσης το earmarking είναι ακόμη ένας από τους τομείς όπου υποστηρίζουμε φιλόδοξες θέσεις και προτιμούμε το shall σαν διατύπωση παρά το should. Το πρόκειται να και όχι το θα έπρεπε. Θέλουμε δηλαδή να είμαστε πιο φιλόδοξοι πάντα. Η ρήτρα ότι ο Ριπένον πληρώνει παραμένει ζήτημα δυσαρέσκειας, δεν είναι ικανοποιητική δηλαδή η ε, λύση που έχει δοθεί. Υπάρχει μια πρόταση με τέλη στις περιοχές όπου εμφανίζονται συνήθως οι στην ε, κυκλοφορία μια λύση την οποία εμείς ως ομάδα θα μπορούσαμε να δεχθούμε εφόσον όμως είναι ουδέτερη δημοσιονομική, δημοσιονομικά. Θα πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό θα μπορέσουμε χάρη στις προτάσεις αυτές να επηρεάσουμε τις θέσεις του Συμβουλίου. Είπατε βεβαίως και εσείς και έχετε δίκαιο ότι είναι περιορισμένο το περιθώριο κινήσεως, κινητικότητας. Στο δε τομέα, στο δε πεδίο εφαρμογής προτείνεται ένα πεδίο εφαρμογής ε, στο 3,5% οι Γερμανοί ε, συνάδελφοι δεν έχουν λόγο ανησυχίας δεδομένου των όσων ισχύουν στο γερμανικό σύστημα. Άρα δεν υπάρχει θέμα εκεί. Μετά ανανέωση του στόλου τροπολογία 31 συγκεκριμένα, όταν εδώ ε, υπάρχουν ε, εξαιρέσεις, θα πρέπει ή τα έσοδα να πηγαίνουν στον τομέα προτιμήσεως όπως έχουμε ορίσει. Αυτό το βρίσκουμε πολύ σημαντικό. Το 3% λιγότερο δεν είναι από ό,τι φαίνεται πρόβλημα για τους συναδέλφους. Μπορούμε να δεχθούμε τη δική σας ε, θέση. Επίσης μπορούμε να σας υποστηρίξουμε αύριο στην... Ε, μπορούν να σας υποστηρίξουν κάποιοι συνάδελφοι ίσως να απόσχουν, αλλά εμείς εν γέννη μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στην αυριανή ψηφοφορία. Όπως είπα, η εν γέννη κατεύθυνση που έχετε επιλέξει ε, σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο μας φαίνεται σωστή. Για τη ρήτρα αναθεώρησης. Ζητούμε αναθεώρηση στα 2, 3 ή 5 χρόνια και δεν ξέρω εάν θεωρείτε και εσείς σκόπιμο να ορίσουμε συνθήκες που επιτρέπουν την άμεση εφαρμογή της οδηγίας ε, σε όλα τα κράτη-μέλη, το ταχύτερο δυνατό. Και επομένω, ίσω θα ήταν σκόπιμο να προσπαθήσουμε όχι να πιέσουμε τόσο πολύ τα κράτη-μέλη στο θέμα αυτό, αλλά να τα ε, πείσουμε να δεχθούν την εφαρμογή. Κύριο Στέρξ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές γιατί πιστεύω ότι έχουμε συγκλίνουμε στις θέσεις μας, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αυτό που θα κάνουμε αύριο, δίνουμε χώρο για διαπραγμάτευση στον εισηγητή για να αναφερθεί στο Συμβούλιο. Και κατά τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να ε, έχουμε κάτι το οποίο θα υπερψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Είναι δύσκολο, θα είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις. Εάν πάμε στην ε, συνδιαλλαγή θα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε μια σαφή θέση. Μπορούμε να το κάνουμε, το είπε και ο ίδιος ο εισηγητής και μετά αυτός μπορεί να διαπραγματευτεί. Επίσης πιστεύω και συμφωνώ με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να είμαστε όσο πιο αποτελεσματικοί μπορούμε. Ο ίδιος λέει ότι υπάρχουν κάποιες τροπολογίες με τις οποίες θα συμφωνούσε αλλά δεν ε, θα τις υποστηρίξει γιατί δεν πρέπει να υπερφορτώσουμε ε, το πρόγραμμα αν θέλουμε να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο και συμφωνώ με αυτόν. Υπάρχουν μεμονωμένες τροπολογίες με, το, με τις οποίες θα συμφωνούσαμε, αλλά δεν θα τις ψηφίσουμε διότι αυτό, όπως είπα, βαριφορτώνει το πρόγραμμα. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια θέση που θα μας επιτρέψει να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο σε θέματα αρχής. Πρώτον, η εσωτερικεύση των εξωτερικών ε, δαπανών, τι θέλουμε. Θα μπορούμε να συμφωνήσουμε με του συμβιβασμού και, και χαίρομαι ότι αυτό ε, έχει συνδεθεί και σε άρθρο. Υπήρχε ε, η τροπολογία 94 από την ΕΒΑ, την υποστήριξε και ο εισηγητής. Τώρα για το θέμα του earmarking, του προσδιορισμού, Πιστεύω ότι έχουμε κάνει μια καλή πρόταση. Θα είναι σκληρή συζήτηση με το Συμβούλιο γιατί δεν τους ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό. Δεν είναι πολύ ενθουσιώδης. Όσο πιο σαφή είναι στην οδηγία, τόσο πιο λίγα κράτη-μέλη θα την θέλουν. Ε, σε ό,τι αφορά την εμβέλεια υπάρχει ένα πρόβλημα. Ε, το είπαμε, πολλές, το είπαμε για τους 3,5 τόνους. Ε, δεν συμφωνούν όλοι στην ομάδα μου. Σε ό,τι αφορά τα επίπεδα συμφόρησης, ε, ναι, 200% 8 ώρες. Θα δούμε τι θα γίνει με τις διαπραγματεύσεις. Αλλά... Ε, μπορώ να παρακολουθήσω την Κορίν σε αυτό. Θα δούμε πώς θα προκύψουν τα πράγματα μετά τις διαπραγματεύσεις. Ανανέωση του στόλου. Ε, βλέπω την γραμμή σκέψης του εισηγητή, αλλά πρέπει να πω ότι εμείς δείχνουμε κατανόηση λέγοντας ότι θα πρέπει να υποδείξετε ε, στα προγράμματα προτεραιότητας. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται, τι θα προκύψει από την ψηφοφορία και τι άλλες τροπολογίες θα εγκριθούν. Πιστεύω όμως ότι σε αυτή την Επιτροπή αύριο θα πρέπει να έχουμε μια όσο πιο σαφή θέση μπορούμε και τη μεγαλύτερη πλειοψηφία για να πούμε στο Συμβούλιο ορίστε αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου, θα την υποστηρίξουμε, θα τη διαπραγματευτούμε και θα πρέπει να προχωρήσετε προς τη δική μας κατεύθυνση. Εάν δεν έχουμε μια σαφή θέση θα είναι δύσκολα τα πράγματα και δεν θα πετύχουμε περισσότερο. Για τους πράσινους, η κυρία Ευχαριστώ πολύ. Φαντάζεστε ότι η καρδιά μου στάζει αίμα για αυτές τις διαπραγματεύσεις και ότι πραγματικά δεν, λυπούμε βαθύτατα που δεν προχωρούμε περισσότερο. Προκαταβολικά θα ήθελα να πω ότι όλες οι τροπολογίες, οι συμβαστικές καλύτερα τροπολογίες του εισηγητή για μένα είναι ικανοποιητικές, θα τις υποστήριζα δηλαδή για τον απλούστατο λόγο ότι Εάν ε, τι καταψηφίζαμε, η εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστου, θα χάνονταν τελείω από το παιχνίδι. Για λόγου δηλαδή τακτική περισσότερο θα τι δεχόμουν. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε όμως κάποια στιγμή όχι μόνο το λόμπι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά επίσης να αντιληφθούμε ότι η καρδιά και ο πυρήνα των λόμπι δεν είναι στο Συμβούλιο. Διότι τα προβλήματα, οι ανησυχίες των περί αυτοκίνητων δρόμων έχουν μηδενική αξία, μηδενική, τίποτε περισσότερο από το μηδέν. Και γι' αυτό καλό θα ήταν κάποια στιγμή να δώσουμε χρόνο για μια συζήτηση για τα λόμπι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα για να φερθώ κατευθείαν στις ε, τροπολογίες. Εμφανίζεται ένα πρόβλημα ουσίας, θεμελιώδες μάλλον, ως προς το θέμα της βασικής ιδέας της ε, αποδοχής τέλους για, τους, ε, για τις συμφόρηση στους δρόμους. Ότι δηλαδή θα μπορέσει αυτό να αποτελέσει αυτομάτως ένα αποδεκτό μέτρο και ένα ε, μέτρο marketing λίγο πολύ για την αποσυμφόρηση των δρόμων. Αλλά αυτό προφανώς ήταν λάθος υπολογισμός. Τέλος πάντων, πάει αυτό, ας μην ε, το συζητάμε περισσότερο. Και βλέπουμε ότι έχει χαθεί και αυτή η ιδέα για την συμφόρηση, αλλά και η ιδέα της ε, ευελιξίας στην επιλογή των οδών. Και ο υπολογισμός, ο οποίος θα πρέπει να ενημερώνεται κάθε τόσο, αποδεικνύεται μάλλον δύσκολος και άρα δεν θα είναι καθόλου χρήσιμος. Για το κόστος, ποιος θα επιβαρύνεται με το κόστος. Πάλι τα κράτη-μέλη πιέζουν ιδιαίτερα. Οι 12 ω λύση βλέπουμε ότι θα έχουν μάλλον αρνητική επίδραση, διότι σε τελευταία ανάλυση θα οδηγήσουν στην ε, διάλυση του φορτίου σε μικρότερα φορτηγά και μεταφορά του σε περισσότερα μικρότερα φορτηγά. Η εξωτερήκευση του ιστορικού κόστου του ή άλλω βλέπουμε ότι μόνο για το Euro 1 και 2, από ό,τι προβλέπει το Συμβούλιο, μπορεί να αποτελέσει λύση. Και αυτό πρέπει να το ξανακοιτάξουν οι συνάδελφοι, γιατί θα έχει σαν συνέπεια ότι με την θέση εφαρμογή ή με τι μεταβατικέ διατάξει που θα εισαχθούν, θα έχουμε την δυνατότητα εφαρμογή αυτή τη ομοθεσία μόνο όταν υπάρχουν τέτοιου τύπου ε, αυτοκινητόδρομοι. Με το Euro 3 ουσιαστικά περιοριζόμαστε μόνο στην κεντρική Ευρώπη, όπου υπάρχει το καλύτερο επίπεδο αυτοκινητοδρόμων και άρα χάνουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό από την κυκλοφορία. Δεν ελέγχουμε μάλλον ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό από την κυκλοφορία φορτηγών. Ένα και δύο, επίπεδα 1 και 2, γυρω γύρω ένα-δύο, δεν υπάρχουν ουσιαστικά σε μεγάλες αποστάσεις αυτοκινητοδρόμων, μόνο σε βραχίες αποστάσεις μέσα στα κράτη-μέλη και γι' αυτό παρακαλώ σκεφτείτε το πάρα πολύ προσεκτικά. Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε το γύρο 4, παρακαλώ πολύ, αλλά τουλάχιστον να το γύρο 3. Διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα η νομοθεσία που θα εισαγάγουμε. Και αυτό θα ήταν μέγα σφάλμα εκ μέρου τη Επιτροπή Μεταφορών, δηλαδή να εισαγάγει διατάξει οι οποίε θα έχουν ουσιαστική εφαρμογή επουδενή. Η διαλειτουργικότητα είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό για μένα ζήτημα. Θα πρέπει πιστεύω να ρίξουμε μια ματιά πολύ προσεκτική ώστε να μην ε, υποστηρίζουμε μόνο την επιβίωση των παλαιότερων προτύπων, μοντέλων καλύτερα, αλλά να ενθαρρύνουμε την καινοτομία. Καταλαβαίνω βέβαια ότι και ο εισηγητής προσπαθεί όσο το δυνατόν να αποτρέψει λύσεις οι οποίες ε, αποκλίνουν πολύ από τη συμβαστική του γραμμή και καταλαβαίνω και τους λόγους του, αλλά από την άλλη νομίζω ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε ένα μεγαλύτερο περιθώριο χειρισμών σε σχέση με το Συμβούλιο στις διαπραγματεύσεις μας και γνωρίζω από την άλλη ότι έχουμε να προσκρούσουμε πάνω σε ένα τείχος τείχο από μπετόν στο Συμβούλιο. Είναι η θέση τους ε, αμετακίνητη Και από την άλλη ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε σπουδαίοι όταν πρόκειται να κάνουμε μεγάλες διακηρύξεις, 20% περιορισμού των ε, εκπομπών, των ε, επιβλαβών για την κλιματική αλλαγή κτλ. Όλα αυτά τα κάνουμε πολύ καλά. Αλλά όταν έρθει η ώρα να λάβουμε αποφάσεις, καλού κακού δεν κάνουμε τίποτα. Καλού κακού μένουμε αδρανείς. Αυτό όμως είναι ζήτημα αξιοπιστίας. Και αυτό είναι ακριβώς η πρόκληση την οποία έχουμε να αναλάβουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστών τον ε, Σαΐντ Ελ Χαντραουί γιατί τα έχει κάνει όλα με μεγάλη κομψότητα και με πολύ στρατηγικό πνεύμα αντιμετωπίζοντας τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και με στόχο να μπορέσει να βρει μια συμβιβαστική λύση με όλους τους κοιόδη εισηγητέ. Εμεί έχουμε κάπως διαφορετικέ απόψεις Οι διαφορές μας δεν είναι το ευρωσήμα, την ευρωβινιέτα. Οι απόψεις μας φυσικά προσδιορίζονται από τις γεωγραφικές θέσεις των διαφόρων χωρών και επομένως έχουμε την ανάγκη μιας πολύπλοκης αντιμετώπισης, αλλά πιστεύουμε ότι η θέση που θα ψηφίσουμε είναι μια πολύ καλή βάση για τις διαπραγματεύσεις. Εμείς ως σοσιαλιστική ομάδα δεν έχουμε καταθέσει ποτάσεις τροπολογιών. Όπως είπε η κυρία Λίχτεμπεργκερ, η θέση του Συμβουλίου είναι μια συμβιβαστική λύση την οποία εμεί θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Και θα πρέπει να καταλάβουμε πόσο δύσκολο είναι για το Συμβούλιο να αλλάξει την συμβιβαστική αυτή λύση. Αν ανοίξουν και πάλι τους ασκούς του αιώλου, τότε στο Συμβούλιο, τότε το Κοινοβούλιο θα βρεθεί στη μεριά των χαμένων. Σε ό,τι αφορά το όριο των 12 τόνων. για τη συμπερίληψη λοιπόν οχημάτων μέχρι 12 τόνων. Θα θέλαμε να το αφήσουμε στα κράτη-μέλη το κατά πόσο θέλουν να το πράξουν αυτό. Αυτό είναι στο σημείο 10. Και η ανανέωση του στόλου. Νομίζουμε ότι θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει μια ανανέωση σε επίπεδο τριών ετών. Αυτό είναι μια λύση η οποία είναι λογική για τον προσδιορισμό των εσόδων. Είναι διαφορετικέ τώρα οι θέσει των διαφόρων χωρών μελών και αν λάβουμε υπόψη την ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση, οι Υπουργοί Οικονομικών θα θέλανε να αποφύγουν τη χρήση του προσδιορισμού. Οι περισσότεροι στη δική μα ομάδα υποστηρίζουν την ανάγκη να υπάρξει προσδιορισμό, αλλά πρέπει φυσικά να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Οχτώ ομιλητές έχουμε. Αν μπορώ να σα ζητήσω να είσαστε λοιπόν σύντομοι να περιοριστείτε σε δύο λεφτά παρακαλώ. Εννέα ομιλητέ. Δέκα ομιλητέ, έντεκα ομιλητέ. Ε, ακόμα λιγότερο χρόνο έχετε λοιπόν. Αρχίζω με τον κύριο Γκρό Για δύο λεπτά ο Μάξιμου. Σα ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τους σκιώδεις το αποτέλεσμα που πετύχαμε ως Κοινοβούλιο για την επίτευξη της εσωτερικοποίησης του κόστους νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί κανείς να υποστηρίζει ότι ε, εμείς στο Κοινοβούλιο λειτουργούμε μονάχα στον τομέα του ιδεατού και δεν προσπαθούμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα πραγματικότητα. η στόχη είναι πολύ σαφής. όχι απλώς να γίνει πιο... Δεν θέλουμε να επιτύχουμε να είναι πιο ακριβή η κυκλοφορία στους δρόμου, θέλουμε να την κάνουμε ασφαλέστερη. Έχουμε λοιπόν ένα συγκεκριμένο στόχο, όχι απλώς να πληρώνει περισσότερα τα φορτηγά. Θέλουμε όλα αυτά τα στοιχεία, όλα τα έσοδα να χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των υποδομών. Φυσικά η ευκαμψία είναι ένα θέμα που παίζει ρόλο και έχουμε δείξει και στο Συμβούλιο ότι ως Κοινοβούλιο είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε, δεν έχουμε μία θέση η οποία είναι αδιάλεκτη. Ξέρουμε ότι τα θέματα της ευελιξίας για ζητήματα όπως η ανανέωση του στόλου των φορτηγών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει συζήτηση, αλλά θα πρέπει και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να δείξουν ευελιξία. Αλλά όταν μιλάμε για φορτηγά υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των κατηγοριών ευρώ 0 με ευρώ 4. <clears throat> Υπήρξε μια μεγάλη πρόοδο στην τεχνολογία Κάτι το οποίο υποστηρίξαμε και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε με την ψηφοφορία που θα γίνει να έχουμε μια ισχυρή πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να βρεθεί το Συμβούλιο σε μια θέση που να μην μπορεί να πει ότι δεν είναι ρεαλιστικό να δεχτεί κανείς τι προτάσει του Κοινοβουλίου και να ξέρει ότι αν δεν δεχτεί τι θέσει μα δεν θα υπάρξει καμία πρόταση. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν μια στάση η οποία θα είναι ρεαλιστική και μπορούμε να θέσουμε τη σωστή κατεύθυνση ω Κοινοβούλιο. Εγώ θα ήθελα για τα τέσσερα κύρια σημεία να επιτύχουμε μια ευρεία πλειοψηφία ώστε να έχουμε και ένα σαφέ μήνυμα που θα δώσουμε στο Συμβούλιο. Η κυρία Τικάου για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, κύριο Ελχαντράουι για την έκθεσή του. Δούλεψε πολύ σκληρά για αυτήν. Ε, ήμασταν πολύ φιλόδοξοι σε πρώτη ανάγνωση για να δώσουμε μια εντολή όσο πιο δυνατή για τη δεύτερη ανάγνωση. Υποστηρίζω την θέση ορυπαίνων πυρών και την εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους, αλλά λυπούμε για το γεγονός ότι αυτή η εσωτερήκευση και η αρχή αυτή δεν εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη. Άρα πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να είναι το βήμα για το οποίο να αγωνιστούμε και να έχουμε μια κοινή ενιαία αγορά μεταφορών και αναφέρομαι στις οδικές μεταφορές που να σέβεται και το περιβάλλον. Η εφαρμογή της ε, οδηγίας μόνο από ορισμένα κράτη-μέλη θα, θα δημιουργήσει δυσκολία σε άλλα κράτη-μέλη, για παράδειγμα στα ε, κράτη-μέλη της περιφέρειας, για τα οποία η εφαρμογή αυτής της ε, οδηγίας από μόνο ορισμένα κράτη-μέλη της Κεντρικής Ευρώπης θα σημαίνει ε, κάποιο, ε, ε, κάποιους φραγμούς στο κόστος σχετικά με την μετακίνηση των αγαθών. Άρα άλλα κράτη-μέλη δεν θα είναι πια ανταγωνιστικά στις ευρωπαϊκές αγορές, ίσως και τα προϊόντα να είναι πιο ακριβά και δεν θα μπορούν να ανανεώσουν ούτε τους τόλους τους. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είμαι υπέρ τη ε, ανανέωση τη οδηγια μετα μετά από δύο-τρία χρόνια, δηλαδή να μην την αφήσουμε για ε, μεγάλο χρονικό ε, διάστημα. Έχω κάνει μια τροπολογία έτσι ώστε τα έσοδα να χρησιμοποιούνται και για τις ε, σίγουρες θέσεις στάθμευσης. Αυτοί οι οδηγοί δεν μπορούν να τηρούν τις όρους και τις διατάξεις της, του νόμου σχετικά με τις κοινωνικές διατάξεις για, τις, για τους οδικούς μεταφορείς. Και ε, ειδικά στις ώρες εχμής. Υποστηρίζω τη διαλειτουργικότητα, αλλά προσοχή υπάρχουν πολλά κράτη που έχουν ε, φόρο που ε, στηρίζεται στο χρόνο και όχι στην, στην απόσταση. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μάισνερ, δύο λεπτά ή λιγότερο από δύο λεπτά. Θα τα κάνω και με less, Μπράιν, Θα μιλήσω λιγότερο από δύο λεπτά. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή τη φορά είναι πολύ καλή δουλειά. Έχουμε μια εναλλακτική λύση διαφορετική από την αρχική που είχαμε επί τραπέζης. Είναι πολύ σημαντικό ότι μπορούσαμε να προχωρήσουμε έτσι και ιδιαίτερος προσωπικός θα ήθελα να υπογραμμίσω και βέβαια μιλώ μόνο για τη Γερμανία όπου ξέρετε υπάρχει μεγάλη επιφυλεκτικότητα προς την Ευρωβινιέτα ε, πιστεύω το, ε, το earmarking είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι οι πολιτικοί που ασχολούνται ειδικά με τις μεταφορές στη Γερμανία πιστεύω θα το υποστήριζαν ως λύση, οι άλλοι όχι, αλλά πάντως για τις μεταφορές οι ειδικοί οπωσδήποτε γιατί βοηθάει να προχωρήσουμε προς ανανέωση του στόλου. Πάντως πιστεύω ότι θα πρέπει στα δύο χρόνια να ξανακοιτάξουμε αν έχει λειτουργήσει το σύστημα. Να δούμε αν είχε φέρει τα αποτελέσματα που θέλαμε. Και βέβαια τα 3,5 τόνοι ω λύση και ω ε, μέτρα εξαίρεση ε, θα πρέπει να τα δούμε. Νομίζω ότι ήμουν πιο σύντομη από δύο λεπτά έτσι. Ναι, ναι, όντω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Κράμερ δύο λεπτά. Earmarking. Έχω πει ότι ε, δεν, ε, έχω πει ότι δεν καταλαβαίνω ποιο είναι ο ενθουσιασμό για το earmarking. Του ή άλλω είναι τα συν και τα πλήν του Υπουργείου Οικονομικών αυτά. Για την αναθεώρηση στα δύο χρόνια θα πρότεινα. Και επίσης, κυρία Τιτσάου, δεν πρόκειται να γίνει πιο ακριβό το σύστημα. Ε, έχει κατά τέσσερις φορές υψηλότερα διόδια από τη Γερμανία ή η Ελβετία και έχει 0, 5% μόνο συνολικό κόστο. Γιατί, γιατί έχει 0,05% συγγνώμη. Και αυτό διότι έχουν μπορέσει να ενσωματώσουν ε, τη διαφήμιση κτλ. Και, και ως εκ τούτου είναι όλοι κερδισμένοι. Ακριβώ δεν σημαίνει ότι θα είναι ακριβώ το τελικό αποτέλεσμα. Αρκεί να υπάρχει αποτελεσματική εισαγωγή του συστήματο. Και μην ξεχνάμε επίση ότι δεν έχουμε καμία σχέση με α, θεμητό ανταγωνισμό. Η Κίνα έχει διόδια απεριόριστα ε, αναλογικά με το φορτίο που ισχύουν για κάθε είδους όχημα, ιδιωτικό, δημόσιο κτλ. Ισχύει σε όλους τους δρόμους για κάθε ιδιώτη και μη και εάν αυτό επιβαρύνει το σιδηρόδρομο ε, κατά αυτόν τον τρόπο, εάν μπορέσουμε μάλλον να βοηθήσουμε ώστε να μεταφερθούν τα φορτία προς τον αυτοκίνητό, προς τον σιδηρόδρομο ή μη τι άλλο έχουμε κάτι εξασφαλίσει για το κλίμα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για θεμητό ανταγωνισμό όταν ε, το ζητούμενο είναι το κλίμα, οι κλιματικές αλλαγές. Ευχαριστώ, Βαντάλε. Δεν υποβάλαμε τροπολογία στην ομάδα γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστές δεν πλησιάσαμε ποτέ τόσο κοντά σε μια συμφωνία με το Συμβούλιο. Και βέβαια, ε, κύριε Λίχτεμπεργκ, και εμένα στάζει αίμα η καρδιά μου όταν βλέπω αυτό. Ελπίζω να μην ε, εμοραγώ φυσικά, αλλά ε, έχουμε πάρει μια απόφαση. Αλλά πραγματικά θα λυπόμουν πάρα, πάρα πολύ αν φτάναμε σε κενές αποφάσεις και δεν θέλουμε να αφήσουμε τον έλεγχο που έχουμε εδώ. Ας είμαστε ρεαλιστές. Αν δεν πετύχουμε αυτό που θέλουμε, αν δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε, τουλάχιστον να τηρήσουμε αποχή. Διότι αυτό ενισχύει τη θέση του Κοινοβουλίου. Να είμαστε ρεαλιστές και να τηρήσουμε αποχή εάν πραγματικά δεν μπορείτε να υπερψηφίσετε. Διότι είμαστε πάρα πάρα πολύ κοντά σε μια απόφαση. Είναι καλύτερο λοιπόν ε, με αυτόν τον τρόπο. Κύριος Διγκράντες, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομο. <clears throat> έχω, καταθέσει, έχω υπογράψει μάλλον έξι τροπολογίες. Τέσσερις μαζί με μέλη των αντιπροσωπιών για την ε, Ευρώπη, τη Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ελλάδο και Ισπανία. Η κοινή θέση λοιπόν αυτών των τεσσάρων χωρών δεν είναι τυχαία είναι κάτι το οποίο προκύπτει από την, ε, από την πολικότητα περιφέρειας έναντι κέντρου στην Στην Ευρώπη. Είναι ένα θεμητό, ένας θεμητός συνασπισμός συμφερόντων. Γιατί αυτές οι ρυθμίσεις ευνοούν κάποιους αλλά θίγουν κάποιους άλλους. Γι' αυτό θέλω να κάνω μια σύντομη επισκόπηση των τροπολογιών. Δεν θέλω να σας κουράσω βέβαια γιατί είναι δεδομένη η θέση των περισσότερων σε αυτή την ε, τροπολογία. 52. <clears throat> για τα κίνητρα για την ανανέωση του στόλου και το χρονικό διάστημα της εφαρμογής εξωτερικού κόστους για τα ρηπαίνοντα αυτοκίνητα. Είναι η τροπολογία 52. Από τις κοινέ τροπολογίες 66. Για το φόρο συμφόρησης η τροπολογία μας προτείνει 100% τρίτον. 67 τροπολογία για την εφαρμογή του τέλους συμφόρησης σε σχέση με τις ε, ώρες της ημέρας. Εμείς προτείνουμε τρεις ώρες την ημέρα. Τέταρτον, τροπολογία 102 για το μέγιστο τέλος για ρήπανση. Η τροπολογία μας προτείνει να ε, για ένα χρόνο ακόμα μέχρι το 2018 την κατηγορία ευρώ 6 και έχω καταθέσει και δύο τροπολογίες ο ίδιος προσωπικά. Η πρώτη είναι 63 για την ε, κατανομή κόστους σε ορεινές περιοχές εκτός από τις κατηγορίες οχημάτων Euro 012 και 83 για το προσδιορισμό των τελών. Το Συμβούλιο θέλει αντί να χρησιμοποιήσει το, Συμβούλιο ε, την ε, κατηγορηματική στάση, έχει μια υποθετική στάση. Εμείς ζητάμε τα συνολικά έσοδα να χρησιμοποιηθούν από τα τέλη αυτά, να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση της οδικής υποδομής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι συζητάμε για ένα θέμα εξαιρετικά σοβαρό και στην ουσία του αλλά και στο συμβολισμό του. Ε, και αντίστοιχη σοβαρότητα του θέματος είναι και η εισήγηση του ΣΑΙΔ. Θέλω μονάχα να επισημάνω δύο ζητήματα, κατά τη γνώμη μου ε, κομβικά για και καθοριστικά για την εφαρμογή αλλά και αποτελεσματικότητα αυτού του εργαλείου. Το πρώτο είναι ότι το σύνολο των εσόδων θα πρέπει να διατίθεται για την βελτίωση των υποδομών και το δεύτερο, ε, για την βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα του εργαλείου απαιτείται ε, η υιοθέτησή του από το σύνολο των χωρών μελών. Και αυτό θα πρέπει να είναι, αφού τώρα δεν είναι ρεαλιστικό ο στόχος, θα πρέπει να είναι στόχος μας για την άμεση την πρώτη αναθεώρηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρίκε για δύο λεπτά. Πάρα πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω ευχαριστώ τον Σάιτ και είναι μια μεγάλη πτυχία που προέρχεται από τη Βελγική Προεδρία η διαδικασία αυτού του νομοθετήματος. Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση. Η διαφορά σε προσέγγιση εδώ αφορά, όπως είπε ο κύριος ε, αφορά την διαμάχη μεταξύ των χωρών οι οποίες είναι περιφερειακές με αυτές οι οποίες είναι κεντρικές και οι οποίες υποστηρίζουν την εσωτερικοποίηση του κόστους γιατί προφανώς αυτές επομίζονται το κόστος των υποδομών. Η μεταφορά λοιπόν σε άλλες μορφές Μεταφορά είναι κάτι το οποίο επίση θα πρέπει να το υποστηρίζουμε. Οι διαφορέ μα εδώ δεν ήταν λοιπόν ιδεολογικού χαρακτήρα, είναι πρακτικέ, γι' αυτό πηγαίνουν εγκάσια μέσα από τι πολιτικέ παρατάξει και θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τι προσπάθειες που έκανε για να καταλήξει σε μια συμβαστική λύση. Τελευταία μου παρατήρηση όμως είναι η εξή. Εγώ θα ήθελα να αναρωτηθώ αν έχουμε ενώπιόν μα ένα νέο σύστημα από την πλευρά του Συμβουλίου που συνίσταται στο να, κάνουμε προτά, να κάνει προτάσεις λέγοντας η πλειοψηφία μας είναι επισφαλής, προσέξτε μην την αλλάξετε την πρότασή μας. Αυτό είναι σαν να λέει στο Κοινοβούλιο, προσέξτε, μην αγγίξετε την συμβαστική θέση του Συμβουλίου, δεν θα σπάσει, δεν θα, μην κάνετε τροπολογίες. Και από την άλλη μεριά, εμεί θα πρέπει από τη δική μα πλευρά να έχουμε μια ευρία πλειοψηφία στη θέση του Κοινοβουλίου για να δείξουμε πόσο σημαντική για μα είναι αυτή η τροπολογία. Αυτό δεν, η, η, το νομοθέτημα, Αυτό αφορά και την Ευρωβινιέτα, αλλά σημαίνει το ίδιο και για άλλα νομοθετήματα και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να τονίσουμε τη σημασία του έργου του Κοινοβουλίου μέσα στη συνθήκη της Λισαβόνας. Thank you. Next for two minutes is, uh, Mr. Ο κύριος Πέρκερ. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Μεταφορών, κύριε Πέρκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για αυτά που... για τα καλά σας λόγια. Μαζί με τον κύριο Ρίνκε έχουμε φέρει ορισμένε τροπολογίε. Και εγώ πιστεύω ότι ο εισηγητή έχει ακολουθήσει ένα πάρα πολύ ρεαλιστικό δρόμο και εφόσον πρέπει να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει ένα σαφέ μήνυμα. Τρία σημεία θέλω να δείξω. Πρώτα απ' όλα, όταν εμεί θέλουμε να εξασφαλίσουμε μικρότερε εκπομπέ ρήπων, πρέπει να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο τουλάχιστον δρόμο, που είναι η ανανέωση του στόλου των φορτηγών. Και εδώ χρειάζεται μια παροχή κινήτρων. Οι κατηγορίες 0 έως 2 δεν θα πρέπει να είναι οι μόνες οι οποίες θα καλύπτονται από αυτό το σύστημα. Θα πρέπει να, να επεκτείνουμε το σύστημα των διοδίων και σε άλλες κατηγορίες τουλάχιστον από το 1 ως το 3. Για το λεγόμενο markup, για, την, για το πρόσθετο τέλος για τις ορεινές περιοχές, χρειαζόμαστε εδώ και πιο ε, ευέλικτα εργαλεία, να έχουμε και κάποιες απαλλαγές για να υποστηρίξουμε το στόχο αυτό. Αλλιώς δεν θα είμαστε καθόλου ε, αξιόπιστοι αν επιφέρουμε αυτές τις προσαυξήσεις χωρίς συγχρόνως να δίδουμε και απαλλαγές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και επίσης φυσικά είναι φανερό ότι ο στόχος της συλλογής τελών αυτών θα πρέπει να είναι και η ελάφρυνση στα τέλη των πιο ευαισθητών κατηγοριών οδικών μεταφορέων. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά κύριο Κούν. Πρόεδρε, και εγώ ευχαριστώ τον συγγητή και τους και συγγητές που μπόρεσαν να καταλήξουν μια συμβαστική λύση για μια κοινή θέση του Κοινοβουλίου που θα μας επιτρέψει και ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ιδιαίτερα για τα κράτη διαμετακόμιση στο κέντρο της ε, Ευρώπης, Γερμανία πρώτα απ' όλα. Και επίσης στο κέντρο της Ευρώπης υπάρχουν, ε, όπως ξέρετε, διαφορετικά συστήματα δύο-δύο στα διάφορα κράτη. Και άρα καλό θα ήταν να μην αρχίσουμε να λέμε αυτό το σύστημα που υπάρχει πρέπει να το απαλείψουμε τελείως και να ξεκινήσουμε από το μηδέν, αλλά όπως προτείνεται στην τροπολογία 10, να ορίσουμε ως σημείο υπολογισμού τους 3,5 τόνους και τους 12 και χωρίς να ε, αλλάξουμε ουσιαστικά τα συστήματα να προχωρήσουμε. Για τα δε, υφιστάμενα συστήματα θα πρέπει πιστεύω να τα συνδέσουμε μέσω του συστήματος Γαλιλαίου, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να έχουν πέντε διαφορετικά blue boxes στα φορτηγά όταν περνάνε από διαφορετικά σύνορα από μια χώρα στην άλλη. Και από την άλλη θα πρέπει να διαπιστώσουμε και ότι ε, οι οδικέ μεταφορέ, ιδιαίτερα για τι μικρέ δομέ των επιχειρήσεων που έχουμε, για τι μικρέ επιχειρήσει, ε, ε, είναι πολύ σημαντικά. Και μάλιστα άκουσα σήμερα το πρωί, διάβασα μάλλον στι ειδήσει, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να αυξήσει τα καύσιμα, το φόρο στα καύσιμα κατά 60%. Ρωτώ λοιπόν πώς θα μπορέσουμε τότε να προχωρήσουμε σε ε, ανανέωση του στόλου όταν είναι τόσο ακριβά τα καύσιμα, ειδικά για τι μικρέ επιχειρήσει. Και αυτό δεν χρειάζεται διεξοδικότερη συζήτηση. Ευχαριστώ, Φιτάντσα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον συγητή και τους κοιόδης συγητές ιδιαίτερα την Σκιώδη Σκητρέκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Όπως είπαν οι συνάδελφοι λοιπόν που εξέφρασαν την υποστήριξη τους στις ε, προτάσεις της Ιταλικής αντιπροσωπείας. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία μας δημιουργούν δυσκολίες. Δεν θέλω να τα επαναλάβω και να επανέλθω πολύ σύντομα. ως προς τη διαβάθμιση για την ε, συμφόρηση στους δρόμους, όσον αφορά τις, ε, τα διόδια σε ορισμένες οδούς όσον αφορά τα οχήματα τύπου Euro 6, κατηγορίας Euro 6. Σε όλα αυτά μπορούμε να συμφωνήσουμε και θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουμε καταγράψει μια κοινή θέση, έχουμε υποστηρίξει την κοινή θέση Επίσης συμφωνούμε στην απόσυρση της τροπολογίας υπαριθμών 6 από τον εισηγητή αυτή που έχει να κάνει με τους εναλλακτικού διαδρόμους. Πέραν αυτού ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις και μέσα στις πολιτικές ομάδες. Η πρόταση επίσης ε, νέας διατύπωσης μιας τροπολογίας από την πλευρά των σοσιαλιστών εκεί όπου γίνεται λόγος για παράλληλους ή γειτονικού δρόμους που μπορεί να έχουν ανταγωνιστική λειτουργία. Ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε αν και θα προτιμούσουμε μια διαφορετική διατύπωση. Είπα προς αυτά ως αποτέλεσμα και πραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χίγκιν όμως τώρα, παρακαλώ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ασφαλώς, χωρίς να έχουμε τέτοια έκθεση θα υπάρξουν πάντα και διαφωνίε και συγκρούσεις και τα λοιπά γιατί πρέπει να βρει κανείς τη τομή μεταξύ περιβάλλοντος και οικονομίας και αφετέρου μεταξύ κεντρικών ε, κρατών της, Ευρώπης, και, ε, κρατών της Κεντρικής Ευρώπης και αυτών της περιφέρειας όπως ανέφεραν και η κυρία Τιτσά και ο κύριος ε, Ζήλε νωρίτερα. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε και με πολιτικές αλλά και με οικονομικές ε, ιδέες, μελήματα πολιτικά και οικονομικά που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ιδιαίτερα ορισμένε περιοχέ χρειάζονται ε, κατά τεράστιο βαθμό. Ε, προσωπικά η πατρίδα μου κατά 92% από τι οδηγίε στι δικέ μεταφορέ. Δηλαδή ό,τι κάνουμε, στέλνουμε στην Ευρώπη, στην Αφρική, ό,τι έχει να κάνει με τι οδικέ μεταφορέ. Και οποιαδήποτε επιβάρυνση σημαντική αυτών θα είχε τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις. Πρέπει λοιπόν να πολύ Επίσης, είμαστε όχι μόνο νησιωτική χώρα, αλλά και νησί ε, που είναι παράρτημα ενό άλλου νησιού, περιπτώσει. Είναι κοντά σε ένα άλλο νησί. Και πάλι αυτό σημαίνει επιπλέον δυσκολίε. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι θα πρέπει να συζητήσουμε θέματα όπως αναδιάρθρωση των οδών, όπως σημαίνει ανανέωση του στόλου, όπως είπε η κυρία Τιτσάου νωρίτερα, ε, μελέτη του, του υφασταμένου χώρου της επιφάνειας που υπάρχει στη θέση μας. Όλα αυτά λοιπόν όμως θα καταλήξουν τελικά σε ένα ουσιαστικό οικονομικό πλεονέκτημα. Ποια είναι η επόμενη δηλαδή βαθμίδα που θα μας επιτρέψει να κάνουμε μια επένδυση αποδεδειγμένα χρήσιμη και οικονομική και περιβαλλοντικά ε, αξιοποιήσιμη παραγωγική. Και επίσης, κύριε Λίχτεμπερκ, όλοι θέλουμε να υποστηρίξουμε την πράσινη ατζέντα και όλων μας η καρδιά εμάς, εν πάση περιπτώσει, αλλά ε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε και με το περιβάλλον, αλλά και με ένα πραγματικό κόσμο, με πραγματική οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Πασκουαρέλα, εκ Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας εκ μέρους της Επιτροπής τον εισηγητή και του σκιώδης για το πολύ επικοδομητικό έργο που επιτέλεσαν και που κατέληξε σε μια θέση διαπραγμάτευσης ρεαλιστική απέναντι στο Συμβούλιο που εάν αληθεύει ότι ε, έχει 1,5 χρόνο που έφτασε σε αυτή την κοινή θέση ε, στις πρώτες, στους πρώτους τριμερείς διαλόγους άκουσε το Κοινοβούλιο σε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό τροπολογιών. Αλλά οι συζητήσεις με το Συμβούλιο έχουν επίσης δείξει τον χώρο ε, τον στενό χώρο για ελιγμούς ε, που υπάρχει. ακούσαμε προσοχή τον κύριο Κέλλα, λέω ότι το Συμβούλιο έχει κάνει κάποιες υποχωρήσεις ήδη. Θα ήθελα δεν είναι ο ρόλος της ε, Κομισιόν να βάλει τάξη σε αυτές τις υποθέσεις, αλλά θα ήθελα να επενθυμίσω ότι υπάρχουν κράτη-μέλη που ε, συμφωνούν με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή και ε, θα ήταν και πρόθυμα να υποφεληθούν μια θέση που μπορούσε να οδηγήσει σε αποτυχία της συμφωνίας. Άρα αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δώσουμε ε, να δούμε αν υπάρχει θέση διαπραγμάτευσης. Δεν θα απαντήσω στις διάφορες παρεμβάσεις που ακούστηκαν ε, για την ουσία του θέματος. Θα ήθελα να περιοριστώ σε κάποιες παρατηρήσεις για τις τροπολογίες, ομαδοποιώντας τις σε δύο ομάδες. Πρώτον, οι τροπολογίες για τις οποίες, ε, με τις οποίες συμφωνεί η Κομισιόν και άλλες με τις οποίες δεν συμφωνεί και τόσο πολύ η Επιτροπή. Στην πρώτη κατηγορία των τροπολογιών θα έβαζα αυτές που επιτρέπουν να ε, διασφαλίσουν σε περίπτωση διαβάθμισης το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να οδηγήσει σε ουδετερότητα δημοσιονομική, τροπολογίες που μπορούν να συνδυάσουν την προσάυξηση με την ε, εσωτερικεύση του εξωτερικού κόστους ε, τώρα υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με τις κατηγορίες ε, Euro 0, 1 και 2. Θα πρέπει ακόμη να διαπραγματευτείτε και να βρείτε λύση για τις κατηγορίες 3 ε, καθορίζοντας ενδεχομένως μία ημερομηνία έναρξης, κάποια χρόνια μετά την θέση σε εφαρμογή της ε, οδηγίας για την Ευρωβινιέτα. Το Κοινοβούλιο όμως δεν πρέπει να επιμείνει ε, στην ε, Ευρω 4 που δεν έχει πιθανότητες να την αποδεχτεί το Συμβούλιο. Και τέλος οι τροπολογίες με τις οποίες, μάλλον σε αυτές τις τροπολογίες έχουμε και την ε, συμβαστική τροπολογία για τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών διοδίων. Και αντιστοιχεί στο έργο το οποίο κάνει η Επιτροπή αυτή τη στιγμή, η οδηγία του 2004 καθορίζει ε, τις διατάξεις εφαρμογής καθορίζουν ένα χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της λειτουργίας αυτής από το 2012. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει μια έκθεση που ε, αναφέρεται στην πρόοδο που έχει επετελεστεί και ε, οι επιχειρηματίες θα κάνουν ε, διαθέσιμες αυτές τις υπηρεσίες και αυτό είναι ε, στο θέμα της συμβαστικής τροπολογίας. Υπάρχουν όμως και τροπολογίες για τις οποίες η Κομισιόν εκφράζει κάποιε αμφιβολίε. Θα αναφερόμουν στο 70, τροπολογία 71 πρώτα απ' όλα για την διαβάθμιση των ε, διοδίων, για την ε, δημοσίευση ενός μεν εγχειριδίου για αυτή τη διαβάθμιση. Αυτή η διαβάθμιση ήδη υπάρχει σε κράτη-μέλη, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Τσεχία προβλέπεται και στο νόμο για τις παραχωρήσεις στην Ιταλία, τις συμβάσεις στην Ιταλία. Ε, αρκετά κράτη-μέλη δεν έχουν πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις για τη διαβάθμιση του δικτύου και δεν μπορεί η Κομισιόν να δώσει ένα εγχειρίδιο, ένα βαντεμέκουμ. Αλλά αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι αυτή η αρχή της διαβάθμισης ε, της ε, συμφόρησης δεν μπορεί να το δει κανεί ε, ταξίδι προς ταξίδι, επιχειρηματία προς επιχειρηματία, αλλά θα πρέπει να το δούμε σφαιρικά για ολόκληρο το δίκτυο του κάθε κράτους μέλους και με μια περίοδο αναφοράς των δύο ετών που αναφέρεται στο σημερινό κείμενο της κοινή θέσης. Στο θέμα της διαβάθμισης αναφέρεται η αύξηση μέχρι το 200%. Ε, είναι νόμιμη αυτή η απέτηση, αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το 175% που έχει προσδιοριστεί στην κοινή θέση 175% της μέγιστης επιβάρυνσης αντιστοιχεί στο 500% που είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο σε σχέση με την ελάχιστη επιβάρυνση στην πρώτη ανάγνωση. 175 ίσον 500. Αυτό που είχατε ζητήσει στην πρώτη ανάγνωση. Δεν χρειάζεται λοιπόν να πάμε παραπέρα. Βέβαια το θέμα το πιο επίμαχο πολιτικός είναι εκείνο του earmarking, του προσδιορισμού των κονδυλίων. Το Κοινοβούλιο ξαναβλέπει τις τροπολογίες πρώτης ανάγνωσης. Είμαστε όμως στη δεύτερη ανάγνωση τώρα. Άρα θα πρέπει να βρούμε κάποια συμφωνία σε αυτό το σημείο. Αυτό που έχει σημασία είναι να υποδείξουμε, και έχω τελειώσει, έχω ολοκληρώσει σχεδόν, ε, να υποδείξουμε διαφάνεια, λογοδοσία από πλευράς των κρατών μελών. Πρέπει να δείξουν πώς θα χρησιμοποιήσουν είτε τα έσοδα των διοδίων, είτε παρόμοια έσοδα για τις επενδύσεις στις μεταφορές. Δεν λέω οδικές μεταφορές, μεταφορές γενικά, ε, με στόχο το πρασίνισμα της Ευρώπης. Και επίσης εδώ έχουμε το μήνυμα της Πράσινης Βίβλου που έχει μόλις δημοσιευτεί από την Κομισιόν όπου παρουσιάζεται ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο σε ό,τι αφορά την εσωτερικεύση του εξωτερικού κόστους. Όχι μόνο για τις οδικές ε, μεταφορές, υπάρχουν ε, συγκεκριμένες δράσεις που έχουν ανακοινωθεί και η Κομισιόν, ο κ. Κάλλας το είπε, θέλει να πάει προς μια ε, υποχρεωτική εσωτερήκευση. Ένα σύστημα διοδίων υποχρεωτικό κο για όλους τους χρήστες των μέσων μεταφοράς. Αλλά όλα αυτά δεν θα γίνουν εφικτά αν δεν έχουμε μία συμφωνία για την Ευρωβινιέτα. Η συμφωνία αυτή είναι το κλειδί για να δώσουμε τη δυνατότητα στην Κομισιόν να ακολουθήσει το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριε Αλκαντράου, θέλετε να πείτε κάτι εν συντομία. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομος θα είμαι να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους συναδέλφους μου για την υποστήριξη που μου έχουν δώσει. Πιστεύω σε γενικές γραμμές ότι το πακέτο στο οποίο συμφωνήσαμε μεταξύ σκιωδών εισηγητών και μου του ίδιου θα υποστηριχθεί <clears throat> από την ευρεία πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής μας και για μένα είναι μια ισορροπημένη δέσμη προτάσεων. Όλοι έχουν κάνει παραχωρήσεις και αύριο μπορούμε να δώσουμε ένα στεναρό μήνυμα ότι έχουμε μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση και θα πρέπει με αυτή να βελτιώσουμε και τη θέση του Συμβουλίου. Προς την Κομισιόν. Εμείς έχουμε δεχτεί 90% της θέσης του Συμβουλίου. Γιατί δεν καταθέσαμε για αυτό το κομμάτι τροπολογίες. Δείξαμε ότι είμαστε ευέλικτοι. Αλλά υπάρχουν κάποια θέματα που είναι πολύ σημαντικά για μας. Το earmarking, ο προσδιορισμός είναι ένα από αυτά. και ξέρουμε ότι θα πρέπει και στον τομέα αυτό να καταλήξουμε σε μια συμβαστική θέση. Είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Αλλά όχι τη θέση του Συμβουλίου ως έχει. Πρέπει να είναι συμβαστική. Πρέπει και από τις δύο πλευρές να γίνουν παραχωρήσεις. Όχι απλώς να δεχτούμε μηχανιστικά αυτά που λέει το Συμβούλιο. Ελπίζω ότι το μήνυμα αυτό λοιπόν θα φτάσει στο Συμβούλιο. Και τέλος να πω κάτι για τον ε, ουσιαστικό αντίκτυπο στην πράξη. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ανησυχούν για την ανταγωνιστικότητα. Ναι, θα υπάρξουν ίσως προβλήματα, αλλά θα πρέπει να ανταγωνίσουν ότι η αύξηση της τιμής του δίζελ στους πρόσφατους μήνες και στο μέλλον, και στο μέλλον θα έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο σε ό,τι αφορά το κόστος από τη μικρή ενδεχόμενη αύξηση στα διόδια επί τη βάση αυτής της οδηγίας. Θα είναι μονάχα μερικά λεπτά του ευρώ ανά χιλιόμετρο και όχι παραπάνω. Ενώ η αύξηση του διζελ είναι πολύ μεγαλύτερη τη τιμή του ντίζελ. Υπάρχει μια άλλη μεγάλη <coughs> σημαντική διαφορά. Η τιμή του διζελ είναι για όλους η ίδια. Αλλά η οδηγία αυτή επιτρέπει στους μεταφορείς να αποφύγουν κάποιες μορφές κόστους, γιατί ένα νέο φορτηγό επιβαρύνεται λιγότερο από άλλα φορτηγά. Αν αποφύγετε τις ε, περιόδους, τις ώρες εχμής στο δρόμο πληρώνεται λιγότερο πάλι. Υπάρχει αυτή η διαμόρφωση λοιπόν. Πάση περιπτώσει μπορώ να σταματήσω εδώ και ελπίζω θα, τα... θα συμφωνήσουμε στην ψηφοφορία αύριο. Ναι, η ψηφοφορία προβλέπεται για αύριο το πρωί και η Ολομέλεια, στην Ολομέλεια θα έρθει το θέμα αυτό τον Ιούνιο. Σας ευχαριστώ. Το επόμενο θέμα είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής με εισηγητή τον κύριο Κουμουτσάκο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, αναφέρατε, θα περιμένω λίγο να βγουν οι συνάδελφοι που δεν ενδιαφέρονται από την ε, ενιαία θαλάσσια πολιτική. Σας παρακαλώ να αποχωρήσετε ηρέμους, ησύχως και ταχαίως, λέει ο πρόεδρος στους βουλευτές που φεύγουν. Ευχαριστώ. Για κύριε αν θέλετε. Όπως ε, ήδη αναφέρατε αύριο ψηφίζουμε τον πρώτο χρηματοδοτικό κανονισμό για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γνωστό κύριε Πρόεδρε ότι το προβλεπόμενο από το σχέδιο κανονισμού ε, ποσών των 50 εκατομμυρίων ευρώ είναι ένα μάλλον μετριοπαθές ποσών. Όμως η ουσιαστική πολιτική σημασία αυτού του κανονισμού για την περαιτέρω ανάπτυξη της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, αυτή της νέας πολιτικής που όλοι έχουμε υποστηρίξει, είναι σημαντική. Σε αυτό το στάδιο πρέπει λοιπόν να επιτύχουμε, προκειμένου στη συνέχεια, όπως προτείνω και με, τις, με συγκεκριμένη τροπολογία, να συμπεριληφθεί η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2014-2020. Την σημασία αυτού του κειμένου που ψηφίζουμε αύριο επιβεβαιώνει το μεγάλο ενδιαφέρον που προκάλεσε. Συγκεκριμένα κατατέθηκαν περίπου 240 τροπολογίες ή άλλες συνεισφορές από τους συναδέλφους της ΤΡΑΝ αλλά και από τέσσερις ε, άλλες επιτροπές που κατέθεσαν τη γνώμη τους η Επιτροπή Περιφερειών, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, η Επιτροπή Προϋπολογισμού και η Επιτροπή Αλίας. Σκοπός μου εξ αρχής ήταν να επιτύχω σε αυτό το κείμενο, να επιτευχθούν σε αυτό το κείμενο πέντε στόχοι. Πρώτον, να υποστηριχθεί από όλου αυτό το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Δεύτερον, να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια για το πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Και αυτό με την εξειδίκευση των γενικών και ειδικών στόχων της πολιτικής. Τρίτος στόχος, να αναδειχθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση της εφαρμογής αυτής της πολιτικής, αυτού του προγράμματος. Τέταρτος στόχος, να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή και σε τακτικά διαστήματα, χρονικά διαστήματα ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Κομισιόν για την πορεία του προγράμματος. Πέμπτος στόχος και σημαντικότερος ίσως να διαμορφωθεί από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια στέρεη, ισχυρή διαπραγματευτική βάση, ώστε να μπορέσουμε στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο να επιτύχουμε το μέγιστο των επιδιώξεών μας. Και προβλέπω, ε, κύριε Πρόεδρε, προβλέπω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο δεν θα είναι εύκολες, διότι οι πληροφορίες είναι ότι υπάρχει απόκληση και όσον αφορά το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και όσον αφορά τις delegated acts που προτείνουμε εμείς εδώ. Λοιπόν, στη βάση αυτών των στόχων προσπάθησα να λάβω υπόψη μου το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό τροπολογιών και των ε, συνεισφορών που κατατέθηκαν. Σε αυτή την ε, προσπάθεια συμβιβασμού και σύνθεσης, όμως, υπήρξε ένα απαράβατο όριο, ένα εμπόδιο αν θέλετε. Είναι το όριο που καθορίζει ο ίδιος ο χαρακτήρας, η ίδια η φύση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Είναι μια οριζόντια πολιτική που επιδιώκει όχι να μεταβάλει ήδη υπάρχουσες και ήδη χρηματοδοτούμενες τομεακές πολιτικές, αλλά να τις συντονίσει και να τις συνδέσει λειτουργικά προκειμένου να υπάρξει προστιθέμενη αξία στην εφαρμογή της. Αυτό το όριο ήταν που με έκανε να μην λάβω τελικά υπόψη μου ορισμένες τροπολογίες ή συνεισφορές συναδέλφων που ήταν στην ουσία τους ιδιαίτερα τομεακές και εξειδικευμένες. Πιστέψτε με ότι χρειάστηκε πολλές φορές πολύ shuttle διπλώμαση για να επιτευχθούν οι συμβιβασμοί. Πιστεύω τελικά και κλείνω με αυτό ότι οι 14 συμβιβαστικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί καλύπτουν τη μεγάλη πλειοψηφία και των ανησυχιών και των προβληματισμών των συναδέλφων και ε, βεβαίως προσβλέπω στην ε, αυριανή ψήφισή τους. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συζητητές των άλλων επιτροπών για το, έργο που ε, παρουσίασαν και που υπέβαλαν τις γνώμες τους. Θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδεις συζητητές για, ε, για το ανοιχτό μυαλό και τη διάθεση συνεργασίας ε, που επέδειξαν, αλλά και βέβαια όλους τους άλλους που συνέβαλαν και τους βοηθούς μας που αντάλλαξαν πολλές φορές ε, ε, απόψεις και emails για να μπορέσουμε να βρούμε το κοινό έδαφος, αλλά και βεβαίως τη γραμματεία. Ε, κύριε Πρόεδρε, αυτά ήταν τα γενικά που ήθελα να πω. Αν θα μου, αν θα μου επιτρέψετε, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο-τρία τεχνικά σημεία, ειδικά στον, στον συμβιβασμό νούμερο 2, τον συμβιβασμό B. Εκεί θα δείτε ότι ουσιαστικά υπάρχει μια νέα πρόταση μια νέα παράγραφος που έχει τον τίτλο «Αρχές για την εφαρμογή ε, της πολιτικής». Σε αυτή ουσιαστικά τη νέα παράγραφο προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη μας και να συμπεριλάβουμε πολλές από τις επιμέρους ανησυχίες, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις των συναδέλφων που όμως δεν μπορούσαν να ενταχθούν στο κύριο κείμενο των σκοπών και των στόχων ε, του κανονισμού. Αυτό λοιπόν είναι ένα καινούριο στοιχείο το οποίο έχει βεβαίως κατατεθεί και έχει τεθεί υπόψη των συναδέλφων. Υπάρχουν ε, ε, και τέσσερις ε, προφορικές τροπολογίες που αφορούν την τροπολογία 117 του κυρίου Μιλάνα. Εκεί επειδή στην αρχική του πρόταση δεν υπήρχε μια αναφορά στη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί νομίζω ότι είναι χρήσιμο να προσθεθεί μια σχετική αναφορά και αυτό επιδιώκει αυτή η προφορική τροπολογία. Στην ε, περίπτωση της τροπολογίας 26 ε, της Επιτροπής ε, Περιφερειών αφορά το άρθρο 10 παράγραφο 6 εκεί πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μια, ένα split vote γιατί νομίζω ότι είναι πιο ακριβές έτσι το περιεχόμενο. Τέλος, ακόμα δύο προφορικές τροπολογίες αφορούν το recital 8 όπου έφυγε μία επιπλέον αναφορά στην Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ε, υπάρχουν και αλλού αναφορές και δεν χρειαζόταν μία ακόμα. Και τέλος ε, υπάρχει ένα split vote στην τροπολογία 1 ε, της Επιτροπής του Προϋπολογισμού γιατί δεν χρειάζεται αναφορά σε ουσιαστικά σε αναθεώρηση, είναι ο όρος λάθος, ε, reviewed λέει η συγκεκριμένη ε, τροπολογία, νομίζω ότι ε, μπορεί να δημιουργήσει αυτός ο όρος παρανόηση ως προς το ότι το πρόγραμμα μπορεί να αναθεωρηθεί κατά την πορεία. κύριε Πρόεδρε, αυτά ήθελα να πω εγώ και να κλείσω ευχαριστώντας και πάλι όλους όσους με τη δουλειά τους και την καλή τους επικοδομητική διάθεση συνέβαλαν στο αποτέλεσμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mr. Ο κύριος Μιλάνα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή με τον οποίο συνεργαστήκαμε πολύ στενά τις τελευταίες εβδομάδες. Ήταν πάρα πολύ πολύπλοκο το θέμα αυτό. Είχαμε πολλά στοιχεία να αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο τροπολογιών και είχαμε και κοινή θέση σε πολλά σημεία γιατί οι συμβαστικές προτάσεις τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δική μας ομάδα είναι απόλυτα αποδεκτές και έχουν γίνει και με συνεργασία μας με τον εισηγητή. Θέλω να <clears throat> υπογραμμίσω την ιδέα αυτή ότι η αξία αυτού του κανονισμού προχωράει κατά πολύ πέραν των θεμάτων των 50 εκατομμυρίων ευρώ, του ύψους δηλαδή των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα μήνυμα προς το Κοινοβούλιο ότι αυτή η πολιτική θα πρέπει να συνεχίσει να την χάνει υποστήριξης. Και επομένως και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των προγραμμάτων θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω χρηματοδότησης για να υποστηριχθεί αυτή η πολιτική. Και αυτό ήταν ένα στοιχείο ουσιαστικό. Και επειδή πρόκειται για ένα κανονισμό ο οποίος έχει σαν στόχο να δώσει τους απαραίτητους πόρους, υπήρξε αυτή η δυνατότητα στο άρθρο 2 και στο άρθρο 3 με τις συμβαστικές λύσεις που πετύχαμε να τονιστεί καλύτερα η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι χρειάζεται και κάποιος προβληματισμός σε σχέση με αυτόν τον κανονισμό. Πρέπει τα 57 εκατομμύρια ευρώ να χρησιμοποιηθούν για κάτι. Δεν πρέπει να μείνουν αδρανοί. Θα πρέπει να συμπληρώσουν τα προγράμματα τα οποία ήδη είναι σε εξέλιξη. Και νομίζω ότι είναι σωστή η ιδέα του Κοινοβουλίου να προσπαθήσει να εξασφαλίσει ότι θα έχουν τη σωστή χρησιμοποίηση αυτά τα κονδύλια. Και είναι σημαντικός αυτός ο κανονισμός γιατί με τον τρόπο αυτό θα βρούμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε την πολιτική μας και να την επικαιροποιήσουμε. Έχει λοιπόν ο εισηγητής απόλυτα την υποστήριξή μου στα θέματα αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κουμουτσάκα. Και σε σχέση με την τροπολογία 117 που είναι πάρα πολύ πολύπλοκο το θέμα που καλύπτει και εγώ υποστηρίζω την θέση αυτή που ανέφερα. Πιστεύω ότι αύριο και η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα μπορέσει να υποστηρίξει πλήρως όλα τα σημεία ε, συμβιβασμού, ακόμα και αν η αρχική μας θέση φυσικά ήταν διαφορετική. Κύριε Μάσνα, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τον κύριο Κουμουτσάκο. Στις διαπραγματεύσεις αυτή της έκθεσης είδαμε ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός συνένεσης. Στην προηγούμενη έκθεση την οποία είχα εγώ αναλάβει στο παρελθόν <clears throat> ήταν ο κύριος Κουμουτσάκος σχεδόν εισηγητής και επομένως είχαμε ένα κοινό μήκο κύματο σε πολλά σημεία. Εμείς δεχόμαστε όλες τις συμβαστικές λύσεις. Αυτό είναι πολύ θετικό λοιπόν γιατί δεν υπήρξε με, δεν υπήρξε ουσιαστική διαμάχη σε σχέση με αυτή την ε, έκθεση. Ξέρετε κύριε Πρόεδρε ότι εγώ υποστηρίζω ιδιαίτερα την ανάγκη να υπάρξει μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και ελπίζω ότι αυτή η πολιτική θα πάρει και μια μεγαλύτερη σημασία. Όλοι οι στόχοι που έθεσε ο κύριος Κουμουτσάκος αξίζουν την υποστήριξη. Τώρα, για τα 57 εκατομμύρια θα πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη χρησιμοποίηση αυτών των ποσών και προφανώς τα 50 εκατομμύρια δεν θα πρέπει να χαθούν, δεν θα πρέπει να τα διαγράψουμε κάπου. Και είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τύχει πλήρους πληροφόρηση και να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία των κατεχώρησης πράξεων delegated acts στην περίπτωση αυτή. Για τις συγκεκριμένες τροπολογίες, πιστεύω όπως είπε και ο κύριος Κουμουτσάκος, ότι ορισμένε από αυτέ τι τροπολογίε μεταφέρουν τα στοιχεία τα οποία υπήρχαν και στην προηγούμενη έκθεσή μου για την ολοκληρωμένη ε, θαλάσσια πολιτική, γιατί έχουν σαν στόχο να εξασφαλίσουμε μια κοινή πολιτική που θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην, από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 50 αυτά εκατομμύρια στα οποία αναφέρομαι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουμε νέου κινητήρε. Ε, πλοίων, για να έχουμε καλύτερη χρηματοδότηση των ενεργειών των ακτοπλοϊκών ε, δυνάμεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα για να έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία και μεγαλύτερη καινοτομία στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής. Αυτός που θα πρέπει να είναι και ο στόχος μας. <clears throat> Και θα πρέπει φυσικά να υπάρξει και ταχεία χρησιμοποίηση αυτών των 50 εκατομμυρίων. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι δεν υπάρχει σημείο διαμάχης και μπορούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στη ψηφοφορία αύριο. Κύριος Τέιλορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς πρέπει να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή, πολύ επικοδομητικός χειρισμός των διαπραγματεύσεων. Τον ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν, μέρος των Πρασίνων για τις εισηγήσεις που έχουν τώρα συμπεριληφθεί στις τροπολογίες. Γενικώ ε, θα συμφωνούσαμε με το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης και τις περισσότερους συμβιβασμούς, παρόλο που αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου μάλλον δεν θα επιτευχθεί συμφωνία. Αλλά ε, ένα μέρος αυτών των ε, θεμάτων μπορεί να είναι αποδεκτό είναι, έχει, έχει να κάνει περισσότερο με τη διατύπωση, τη γλώσσα και όχι τις λεπτομέρειες. Γι' αυτό θα ήθελα να υποβάλω τρεις προφορικές τροπολογίες ε, στις, στους συμβιβασμούς. Και έχει να κάνει με, είναι με τη γλώσσα. Έχει να κάνει με τη λέξη growth. Τι σημαίνει growth. Δεν σημαίνει αποτελεσματικότητα, δεν σημαίνει καλύτερη απόδοση, δεν σημαίνει, δεν σημαίνει δύναμη. Σημαίνει περισσότερο. Πιστεύω ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε ε, την αντοχή ε, για να είναι πιο αποτελεσματικός ο τομέας των μεταφορών, για να βελτιώσουμε την απόδοση. Γι' αυτό να ε, βάλουμε μια μικρή τροπολογία για να καταστήσουμε την οικονομική μεγένθηση με την φράση economic resilience, οικονομική αντοχή. Επίσης, ένας άλλος συμβιβασμός H, όπου εκεί αναφέρεται η πρόθεση πρωτοβουλειών για και πάλι αναφέρεται η λέξη growth. Θα πρέπει να το αντικαταστήσουμε με τη λέξη ανθεκτικότητα. Όταν υπάρχει οικονομική κρίση στον τομέα των μεταφορών, στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, αν έχουμε ε, μια πιο ανθεκτική οικονομική προσέγγιση, θα καταφέρουμε να αντεπεξέλθουμε καλύτερα. Και για τον συμβασμό L θα εισηγηθούμε εκεί όπου λέει αηφόρος οικονομική ανάπτυξη, να το αντικαταστήσουμε με, και πάλι με τη λέξη ανθεκτικότητα. Αηφόρος οικονομική ανθεκτικότητα. Ε, και τέλος, ελπίζω να επιτευχθεί συμφωνία σε αυτές τις εισηγήσεις και προτού επιτευχθεί αυτό θα Είμαι πολύ ευγνώμος αν κάποιος κάπου θα μπορούσε να μου εξηγήσει επακριβώς τι σημαίνει μπλε αηφόρος οικονομική <laughs> ανάπτυξη. Έχω κοιτάξει βιβλία, έχω ρωτήσει εμπειρογνώμονες, το έχω ψάξει στο Google. Δεν έχω βρει έναν ορισμό αυτής της φράσης. Θα μου ζητηθεί να ψηφίσω αύριο. Ε, θα μου ζητηθεί να, να ψηφίσω αύριο. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλάβω περί τίνος πρόκειται προτού φτάσουμε στη φάση της ψηφοφορία. Και πολύ σε συνταμία σε, για τα θέματα όπου δεν συμφωνούμε εισαγωγή ενό σχεδίου ανταλλαγής ρήπων λοιπόν, ε, στο θαλάσσιο τομέα ε, δεν έχουμε βρει βελτίωση των κανόνων για τα σκάφη που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία ή ρηπαίνοντα φορτία ή ε, για ε, την ε, απάλψη της ρήπανσης από υπεράχτιες λειτουργίες. Βέβαια θα προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε αυτά τα θέματα σε μελλοντικές φάσεις και το γνωρίζουμε αυτό, μιλάμε για τα 50 εκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές για το τι μπορούμε να ε, πετύχουμε. Κλείνοντας, ε, πρέπει να πω ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι για να πετύχουμε τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι μόνο σε θέματα μεταφορών, αλλά και σε θέματα μείωσης των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα και της προστασίας του περιβάλλοντος. Και ο ίδιος ο εισηγητής αναφέρθηκε στις ευκαιρίες. Την ευκαιρία με αυτό το έγγραφο να χαράξει μια πολιτική κατεύθυνση στο θέμα αυτό επίσης. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το χρόνο. Ευχαριστώ. Θα χρειαστείτε πολύ χρόνο διαβάζοντας πολλές εκθέσεις ε, για πράγματα που δεν ξέρετε. Αν θέλετε να μάθετε τα πάντα για, για αυτά που πρέπει να κληθείτε να ψηφίσετε. Και η Ολομέλεια είναι το κλασικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης. Ο κ. Ε, Βαντάλεν στη συνέχεια. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω τη βαθιά εκτίμηση που τρέφει προ τον εισηγητή. Έκανε πολλές ε, καλές προτάσεις συμβαστικέ. Και θα ήθελα να πω ότι ετοιμάζουμε, θα έλεγα, στολίζουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο με πολλά θέματα τα οποία μας δεν έχουν ακριβώς σχέση με την ουσία μας, με το δικείμενό μας. Μιλάμε για 50 εκατομμύρια που θα πρέπει να κατανεμηθούν για ένα πρόγραμμα και αν κατάλαβα αυτά που λέει ο κύριο Τέιλορ, ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο που ετοιμάζουμε φτάνει μέχρι τον ουρανό χωρί όμω να έχει θεμέλια, χωρί να έχει βάση. Εγώ εν γέννη συμφωνώ με τον εισηγητή. Ίσως να μην ε, τον υποστηρίξουν σε όλα τα, όλα τα μέλη της ομάδας μου, αλλά από ό,τι βλέπω θα ε, δηλώσουν μάλλον αποχή όπου υπάρχει πρόβλημα. Γιατί θέλουμε να προχωρήσει η έκθεση και να τεθεί σε εφαρμογή η νομοθεσία έχω συζητήσει με τον εισηγητή, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την προφορική τροπολογία υπαριθμών στο θέμα 112, στην τροπολογία 112. Είναι ένα πολύ λεπτό για μας θέμα, πολύ ευαίσθητο και δεν θα θέλαμε να ε, δοθούν πρόσθετα χρήματα στις ευρωπαϊκές αποκεντρωμένες υπηρεσίες. προφορική τροπολογία λοιπόν του κ. Κουμουτσάκου για μας είναι δεκτή. Την υποστηρίζουμε διότι έτσι μπορούμε να αποκλείσουμε τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που έχουν στη τελευταία ανάλυση δικές τους γραμμές ε, προς τον προπολογισμό, δικές τους, δικές τους χρηματοδότηση χωριστή. Ακολουθούμε λοιπόν τον εισηγητή. Ίσως να υπάρξουν κάποιες αποχές. Αυτό είναι όλο. Ευχαριστώ κυρία Βίλσο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα προκαταβολικά να υπογραμμίσω ότι η κατάσταση στα ύδατα της Ελλάδας, της Ευρώπης είναι όλο και χειρότερα, χειρότερη. Έχουμε προβλήματα και ως προς την απόρριψη ε, και ως προς την λάθη μετανάστευση. Άρα θέλουμε να έχουμε μια προστασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση του θαλάσσιου οικοσυστήματος όπως και των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει η βιοπικιλότητα στις θάλασσές μας να διαφυλαχθεί για να μπορέσουν να παραμείνουν οι θάλασσες αυτές πηγές τροφής, για να εξασφαλίσετε και το εισόδημα αυτών που ζουν από την ε, θάλασσα. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να ε, αναφερθώ στην ανάγκη το πρόγραμμα για μια ολοκληρωμένη πολιτική για τις θάλασσες να επικεντρώνεται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλασσών αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν είναι αποδεκτό να ε, επιβάλλεται ευρωπαϊκή πολιτική σε ορισμένα κράτη ε, τρίτα δυνάμει του ολοκληρωμένου προγράμματος, τροπολογία 43 δηλαδή. Επίσης, συγκεκριμένα μέτρα στοχευμένα στην πράξη, μέτρα σχετικά με την υπεραλίευση, παρακολούθηση, ε, monitoring, εποπτεία δηλαδή ε, και δίωξη ακόμη των, ε, της παράνομης αλίας, έτσι ώστε να έχουμε στο δυνατόν περισσότερη μείωση των περιττών ή παραλιευμάτων ή παρεπιπτόντων γενικά προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και οικοσυστήματος και προτείνω όπως ακούθηκε και νωρίτερα από τον εκπρόσωπο των Πρασίνων, ε, να λυθεί το θέμα των ε, ε, αντλειών πετρελαίου μέσα στη θάλασσα, που ξέρουμε ότι σημαντικό κίνδυνο μπορεί να προξενήσουν, όπως είδαμε στον κόλπο του Μεξικού. Έχουμε να κάνουμε όλο και, όλο και πιο έντονους κινδύνους Έχουμε να κάνουμε με δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχονται δυνάμει των διατάξεων περί προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και, με, ε, και να ενσωματώνονται σε ένα γενικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών περιβάλλοντος. Ε, η ασφάλεια στην ανοιχτή θάλασσα επίσης είναι ένας τομέας ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει να αποτρέψουμε και τις περιβαλλοντικές καταστροφές, αλλά και επίσης να σώσουμε ζωές χάρη σε συνθήκες καλές ε, υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας στα καράβια ή στο θάλασσο περιβάλλον. Τροπολογίες έχω καταθέσει την 39, 65 και 82, όπου πιστεύω ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε χάρη σε αυτές θάλασσες καθαρές για τις μελλοντικές γενναίες με συνθήκες κοινωνικές εργασίας ε, αποδεκτές χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζουμε τα ψάρια, δεν πρέπει και να παραγνωρίζουμε τον παράγοντα αλλιέα ψαρά. Πρέπει να σώσουμε τόσο τα ψάρια όσο και τους ψαράδες και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν δεκτές αυτές τις τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γκρός. Ευχαριστώ πρόεδρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Να υπενθυμίσω επίσης ότι θέλαμε να είμαστε... Είχαμε διεκδικήσει την ε, ουσιαστική την καθήλυνα αρμοδιότητα για την ε, διατύπωση της έκθεσης. Τα καταφέραμε και ο κύριος Κουμουτσέκος κατάφερε πάνω απ' όλα να έχει πολύ καλό συντονιστικό ρόλο και μεταξύ βέβαια των σκιωδών εισηγητών αλλά και μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων επιτροπών. Είναι πάρα πολύ καλή δουλειά αυτή και νομίζω ότι δεν ε, έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τέτοιο συνδυασμό ε, μέσα σε 400 τροπολογίες κειμένου το οποίο πραγματικά να αντικατοπτρίζει ε, τα μελήματα και τις ανησυχίες των διαφόρων πλευρών. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μπορούμε να έχουμε εδώ μια ολοκληρωμένη πολιτική για τις θάλασσες που απαιτείται και δεν είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολεί μόνο όταν έχουμε φυσικές καταστροφές στις θάλασσες και έχει μεγάλη επικαιρότητα. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλη σημασία εν γέννη και για μας την Επιτροπή των Μεταφορών νομίζω ότι η προσέγγιση είναι πάρα πολύ καλή. Φυσικά χρειάζονται και χρήματα Ελπίζω να μην ε, αμφισβητούνται τα κονδύλια που έχουν προβλεφθεί, δηλαδή η είδηση που μας δόθηκε εδώ να ευσταθεί και να διατηρηθούν ε, αυτά τα ποσά στη χρηματοδότηση. Αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με ποσά τα οποία θα αφορούν συγκεκριμένες περιοχές, ε, παρόχθιες, παραθαλάσσιες κτλ. Αλλά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφορών αυτών περιοχών και πιστεύω ότι η τροπολογία 52 που είναι εκείνη η οποία ιδιαίτερως αναφέρεται σε χαρακτηριστικά κάποιων περιοχών, δηλαδή κυρίως της Μεσογείου, ε, ναι μεν ε, μου φαίνεται συμπαθής ως τροπολογία, αλλά νομίζω ότι αντίστοιχα θα πρέπει να κάνουμε κάτι για όλες τις περιοχές και γι' αυτό θα πρότεινα η τροπολογία αυτή είτε να αποσυρθεί είτε να μην υποστηριχθεί. Αυτό το ε, μπλε σύστημα που ανέφερε ο συνάδελφος από τους πρασίνους να σας εξηγήσω ότι το πράσινο δεν είναι πάντοτε το χρώμα της υγείας. Το γαλάζιο, το μπλε είναι το καθαρό χρώμα και νομίζω ότι θα πρέπει πάντα να το έχετε υπόψη όταν λαμβάνετε θέση σε τέτοια θέματα τη ολοκληρωμένη προστασία των θαλασσών. Κατά τα άλλα, ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να έχουμε πολύ μεγάλη επιτυχία ε, στην ψηφορία αύριο. Σα ευχαριστώ. Προσπαθείτε να πείσετε τους πράσινους ότι το πράσινο είναι, δεν είναι υγι, υγιές χρώμα για το νερό. Κύριε Ντεμέρ, <clears throat> ο κ. Διανέλης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θεωρούμε ότι ο προτινόμενος κανονισμός εξασφαλίζει τελικά 50 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό εξαιρετικά χαμηλό για την ε, υλοποίηση των τόσο φιλόδοξων στόχων μιας τόσο πολύπλευρης και σοβαρής πολιτικής. Όμως, αν έχουμε την κατάλληλη, τη σωστή και αποτελεσματική αξιοποίηση ε, βάζουμε κάποιες βάσεις για την διεκδίκηση σε μακροχρόνια βάση ε, πολύ σημαντικότερων κονδύλιων. Ε, δύο σημειώσεις. Θεωρώ ότι είναι αξιοσημείωτη η παρατήρηση ότι στις περισσότερες συμβιβαστικές τροπολογίες εντάσσονται οι παράκτιες και οι νησιωτικές περιοχές στην καρδιά της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Αυτό αφενός συνάδει βεβαίως με τις επιταγές της συνθήκης της Λισαβόνας Αφετέρου, υιοθετώντα τη αναγνωρίζουμε ότι η ευημερία των νησιωτικών περιοχών της Ευρώπης είναι συνυφασμένη με την αποτελεσματική αλλά και τη βιώσιμη διαχείριση ετερογενών θαλάσσιων δραστηριοτήτων πολλές φορές είναι και αντικρουόμενες και ασύμβατες μεταξύ τους. Μια δεύτερη ε, σημείωση, η τροπολογία, για την, ε, η 88 αν δεν κάνω λάθος, για την ναυτιλία και το ETS, ε, θεωρώ ότι ε, δεν χωρά σε μία έκθεση όπως αυτή για την οποία συζητάμε, όχι μόνο γιατί σε αυτή τη συγκυρία η Επιτροπή όπως και ο IMO εξετάζουν σε πολύ σοβαρή βάση ε, όλα τα ενδεχόμενα για τη μείωση των ε, εκπομπών της ναυτιλίας, αλλά και γιατί η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει το όχημα της διαμόρφωσης της εν λόγω πολιτικής που είναι πολύ σοβαρότερη από το να χωρέσει σε μια τέτοια τροπολογία. Ευχαριστώ. Thank you, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Είναι πολύ δύσκολο να προσπαθήσει κανείς να εξασφαλίσει μια συνοχή σε όλα αυτά τα σημεία, γιατί είναι πάρα πολύ πολύπλοκο το θέμα. Ένα γλωσσικό μονάχα θέμα. Και εμείς ε, ως αγγλόφωνοι πολλές φορές βλέπουμε εδώ πέρα τα αγγλικά και δεν καταλαβαίνουμε μία. Μερικές φορές η αργό που χρησιμοποιείται στα κοινοτικά έγγραφα είναι απίστευτη. Αλλά θα ήθελα και εδώ να θίξω τα εξή σημεία. Γιατί ο εισηγητής έκανε μια πολύ απιστευτη αλλα θα ηθελα και εδω να δειξω τα εξη προσπάθεια για να καταλήξει σε αυτό το αποτέλεσμα. Λένε οι συνάδελφοι ότι έχουμε μονάχα 50 εκατομμύρια ευρώ. 50 εκατομμύρια ευρώ είναι 50 εκατομμύρια ευρώ από την τσέπη του φορολογούμενου. Ζήτησα την Κομισιό να μας δώσει κάποιες λεπτομέρειες για το πώς αυτά τα 50 εκατομμύρια θα πρέπει να δαπανηθούν και μερικοί υποδείξαμε ότι δεν πιστεύαμε ότι αυτά είναι νέα κονδύλια, ότι θα πρέπει να ληφθούν από τον τρέχοντα προϋπολογισμό. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν ε, ε, επιπρόσθετα ποσά στη διάθεσή τους και χρειαζόμαστε κάποιες απαντήσεις. Αν υπάρχει πρόγραμμα θέλουμε να μας υποδείξουν πώς τα 50 εκατομμύρια ευρώ θα δαπανηθούν. Θέλω να ακούσω λοιπόν την απάντηση και την πρόταση της Κομισιόν εδώ και ακριβώς από πού προέρχεται αυτό το πόσο. Ξέρω ότι είναι από την προπολογισμό και την Επιτροπή Αλίας επίσης. Ε, τώρα, η λέξη integrate στα αγγλικά. Ε, μπορεί να μας παραπλανήσει. Ερχόμενοι από νησί, ένα μεγάλο νησί, το Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει ε, μεγάλος συντονισμός που γίνεται ε, σε πολλά θέματα και μπορεί να εσωματωθεί, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε κάτι το οποίο υποδείχθηκε η κυρία Βίλς νομίζω ότι υπάρχουν και τρίτε χώρε εδώ. Η θαλάσσια πολιτική δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα μεμονωμένο κράτο μέλο που έχει ακτές. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, λοιπόν, να μην αρχίσουμε να ε, παρεμβαίνουμε σε διεθνείς ε, συνθήκες και ε, τις οποίες έχουμε ε, συμφωνήσει. Κάποια άλλα σημεία, αν μου επιτρέπετε Πρόεδρε, από την δική μου αντιπροσωπεία δεν υποστηρίζουμε τη χρήση του, του όρου διασυνοριακός ή χωροτακτικός η θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Ε, υποστηρίζουμε την ε, αρχή της επικουρικότητας. Μπορεί κάποιες χώρες να έχουν διαφορετική άποψη που είναι ορθό, αλλά από τη δική μας άποψη ε, δεν συμφωνούμε με αυτό. Και τέλος, κάποια από τα σημεία που έχουν θίχθει. Μιλάμε για καλή συνεργασία στο θέμα του περιβάλλοντος και στις πρακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν για να διασφαλίσουμε ε, για το κατά πόσο υπάρχει υπεραλίευση, ρήπανση, για την απόρριψη των αποβλήτων, ε, πράγματα τα οποία δεν τη χάνουν σωστά του χειρισμού σε ορισμένα κράτη-μέλη. Και αυτά δεν μπορούμε να τα αποδεχτούμε. Και κάποια κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, δουν τις ευθύνε τους, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε εθνικό επίπεδο. Τι πρέπει να κάνουν στα θέματα αυτά. Γενικά λοιπόν υπάρχουν πολλά θετικά σημεία σε αυτή την έκθεση και θα πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά χρειαζόμαστε απαντήσεις από την Κομισιόν για το πώς θα δαπανηθούν αυτά τα κονδύλια και δεν πρέπει να ξεχνούμε το γεγονός ότι υπάρχουν θέματα επικουρικότητας εδώ και επίσης ότι θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δουλεύουμε επικοδομητικά και ότι υπάρχει διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο προχωρούμε. Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ο κράμα. Ζήτησα το λόγο άλλη φορά γιατί το θέμα αυτό με τα 50 εκατομμύρια των Ευρωπαίων φορολογουμένων βακοσύνολτρα, φυσικά και είναι του Ευρωπαίου φορολογουμένου τα εκατομμύρια αυτά. 50 εκατομμύρια όμως για υποδομές, για το περιβάλλον, για, τις, για οικολογικές θαλάσσιες μεταφορές είναι peanuts όπως λέμε, είναι ψίχουλα. Ας κάνουμε μια αναλογική θεώρηση της κατάστασης, ε, κυρία Φώστερ. οι αεροπορικές μεταφορές που δεν πληρώνουν ούτε φόρο ορυκτού καυσίμου, ούτε ε, ΦΠΑ και έχουν ε, επιπτώσεις σοβαρές από τη στρατόσφαιρα μέχρι το έδαφος με 30 δισεκατομμύρια ευρώ για να μπορούν να παίρνουν τα μεγάλα πριμ όλοι αυτοί οι μάνατζερ των αεροπορικών εταιρεών και σας φέρονται πολλά τα 50 εκατομμύρια για να βοηθήσουμε λίγο το περιβάλλον των θαλασσών. Ξαφνικά θυμάστε κυρία Φώστερ ότι είναι χρήματα του Ευρωπαίου φορολογμένου, μα είναι ψίχουλα. Ψίχουλα αν δούμε την αναλογία. Ευχαριστώ, μα θέλετε να κάτσουμε να τα συζητήσουμε όλα. Και τότε να σβήσουμε τα δισεκατομμύρια του Ευρωπαίου φορολογουμένου που δίνονται κάθε χρόνο σε μεταφορές. Πολύ ευχαρίστω. Ευχαριστώ, λέω Η κυρία Μπενίν, εκ μέρους Επιτροπής. Ένα λεπτό, με συγχωρείτε. Μάισνερ, είπατε κυρία Μάισνερ ότι θέλετε και εσείς το λόγο. Μάλιστα. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι σημαίνει sustainable growth and jobs ε, στη συναδελφό. Δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Εάν σκεφτούμε ότι 30% του πλανήτη είναι στερεά και 70% νερό, θάλασσα, καταλαβαίνετε τι λάθος έχουμε κάνει που έχουμε ρίξει το βάρος στην ε, στη στεριά και όχι στη θάλασσα, στο νερό. Ε, αυτό πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια προβλήματα, τα ίδια σφάλματα και να δώσουμε στο γαλάζιο το δυναμικό του και μια οικολογική δυνατότητα ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ολοκληρωμένη πολιτική για τι θάλασσε. Αυτό σημαίνει blue sustainable ε, growth and jobs. Γαλάζια και βιώσιμη ανάπτυξη και θέση εργασία. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Μπενίνγκ από την Επιτροπή. Ναι, άμα τα καταφέρετε να δώσετε την ατάκα μετά από αυτά που υπόθηκαν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γιατί εμείς προτείναμε αυτό τον κανονισμό στην Κομισιόν. Γιατί θέλουμε... Θέλαμε να υποστηρίξουμε τις δράσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλούς ε, Μήνε και να εξασφαλίσουμε ότι μέσα στι τωρινέ δημοσιονομικέ προοπτικέ θα ευδοκιμήσουν. Ποιε είναι τώρα αυτέ οι δράσει. σας έχουν πληροφορήσει βεβαίω. παίρνετε ετήσιες εκθέσει για την εφαρμογή του. οι τελευταίε ήταν το Μάιο του 2010 και θα πάρετε και άλλε το Μάιο στα πλαίσια του τρέχοντος οικονομικού έτους. Τρεις είναι οι βασικές δράσεις που εστιάζουν σε ενέργειες οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν διατομεακή ανάπτυξη. Μιλάμε για καλύτερη χωροταξία στο θαλάσσιο χώρο καταρχήν, λαμβάνοντας υπόψη την πολλαπλότητα και πολυπλοκότητα των συμφερόντων και εδώ παίζει μεγάλο ρόλο η επικουρικότητα γιατί δεν θέλουμε να αποσύρουμε εξουσίες, να αφαιρέσουμε εξουσίες από τα κράτη-μέλη. Θέλουμε όμως να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη με μια κοινή προσέγγιση να έχουν καλύτερη σχεδίαση. Δεύτερος τομέας είναι η γνώση για τη θάλασσα, να γνωρίσουμε καλύτερα για τα θαλάσσια θέματα και αυτές οι γνώσεις να είναι διαθέσιμες σε όλους και να μπορούμε να προχωρήσουμε στην καινοτομία χωρίς να επαναλάβουμε τα ασφάλματα που είχαμε κάνει με άλλους φυσικούς πόρους και τέλος ολοκλήρωση της θαλάσσιας εποπτείας, το οποίο σημαίνει ότι τα τωρινά συστήματα εποπτείας και παρακολούθησης είναι διασυνδεδεμένα και μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε όλοι με λιγότερα χρήματα. Ουσιαστικά καλύπτουμε τα χάσματα μεταξύ διαφορετικών κατατομής πολιτικών στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Γι' αυτό χαιρετίζουμε τις τροπολογίες σας και ιδίως το έργο του εισηγητή με στόχο να υπάρξει αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης και να εξασφαλίσουμε μια συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφορών δράσεων. Δεν θέλουμε να υποστηρίξουμε κατατομής πολιτικές, απλώς να εξασφαλίσουμε ότι εντοπίζουμε τα σημεία συναρμογής μεταξύ των τομιακών πολιτικών για να έχουμε την καλύτερη και πιο εποφελή λειτουργικότητά τους. Εμείς δεν θέλουμε για αυτό το λόγο να έχουμε και άλλες δράσεις και να πολλαπλασιάσουμε τους ε, στόχους, γιατί ο στόχος μας δεν είναι να έχουμε μια κεντρική πολιτική, αλλά να, ο στόχος είναι να λειτουργήσουμε καλύτερα σε μια συνεκτική πολιτική. Μόνο, 30, μόνο τρία χρόνια μας μένουν μέχρι το, μέχρι το τέλος του 2013 και 50 εκατομμύρια θα έχουμε αν συμφωνήσει και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο στόχος λοιπόν να συνεχίσουμε τις προσπαθίες μας, θα συνεχίσουμε να σας δίνουμε πλήρες εκθέσεις για τα θέματα αυτά και στις εκθέσεις αυτές θέλουμε να δείξουμε πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις συγκεκριμένες αυτές δράσεις και να επηρεάσουμε ένα ευρύτερο πεδίο πολιτικών. Αυτό είναι ακριβώς που κάνει και η Κομισιόν <clears throat> με την, ε, με, το, με κυρία Δαμανάκη και τις ομάδες εργασίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κουμουτσάκος, αν θέλει να προσθέσει κάτι. Uh, Πάρα πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, να σας ε, επαναλάβω ότι η δική μας κατανόηση δεν είναι να αλλάξουμε πολιτική, αλλά να γεφυρώσουμε διάφορους τομείς πολιτικής και να δημιουργήσουμε συνέργειες μεταξύ διαφορετικών τομεακών πολιτικών. Δεν μπορώ να συμφωνήσω για αυτό το λόγο με κάποιες από τις τροπολογίες των Πρασίνων και του κυρίου Τέιλορ και γι' αυτό έχουμε καταλήξει σε, στη συγκεκριμένη θέση που σας παρουσιάσω. Για την ε, προσθήκη της ανθεκτικότητας, μάλλον για την αντικατάσταση της ανάπτυξης με ανθεκτικότητα, εγώ δυσκολεύομαι να καταλάβω τι ακριβώς είναι η ανθεκτικότητα. Έχω ελέγξει τι λέει το λεξικό και λέει ότι η ανθεκτικότητα, resilience, είναι η ικανότητα ενό υλικού να επανέλθει στο αρχικό του σχήμα ή στην αρχική του σύσταση όταν έχει υποστεί ε, εντάσεις. Είναι ουσιαστικά μια μορφή ευκαμψίας. Αν θέλει ο κύριο Τέιλερ μπορούμε να μιλήσουμε για ευκαμψία και όχι για ανθεκτικότητα. Και εγώ έχω προβλήματα με την ε, ορολογία και απαντώ εδώ στην κυρία Φώστερ η αργό που χρησιμοποιούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυσκολεύει το ΑΡΓΟ όλων μας, <clears throat> αλλά πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να είναι γενικά αποδεκτό από τους περισσότερους συναδέλφους και φυσικά η συζήτηση για το ολοκληρωμένο, το integrated. Ίσως είναι θεολογικού χαρακτήρα η συζήτηση στο θέμα αυτό. γιατί αν δεχόμασταν την τροπολογία για το ολοκληρωμένο, εγώ θα έπρεπε να αλλάξω τον τίτλο της πολιτικής. Και αυτή ήταν μια δυσκολία που δεν μπορούσα εγώ να ξεπεράσω. Και γενικά σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και την υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Τέιλορ, θέλετε να επανέλθετε. Δεν είναι το πώς ορίζουμε τα χρώματα στο ουρανιοτόξο, είναι κάποιο άλλο θέμα, δεν είναι χρωματικό. Όχι, Πρόεδρε. Απλώς θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και φυσικά έχουμε θεμελιώδεις διαφορές. Είναι διαφορετική η ανάπτυξη και η ικανότητα ανάκτησης, στη resilience, η ανατεκτικότητα είναι διαφορετική. Αλλά θα δούμε τι θα προκύψει από την ψηφοφορία. Ξέχασα όμως να πω κάτι. Και αυτό είναι ότι σε πνεύμα συνεργασίας πράγματι αποσύρουμε τις τροπολογίες 68 και 76 και αν μπορείτε να δείξετε λίγη ευκαμψία κύριε Κουμουτσάκο στην αυριανή ψηφοφορία θα σας είμαστε ευγνώμονες. Ωραία. Ψηφοφορία αύριο και στην Ολομέλεια θα πάμε τον Ιούνιο. Ξεχνάτε πράγματα κύριε Τέιλορ. Αυτό είναι όταν προσπαθείτε να διαβάσετε τι θα ψηφίσετε και τι δεν θα ψηφίσετε, λέει ο πρόεδρος. Στη συνέχεια, τουρισμός στην Ευρώπη. Ο κύριος Φιντάντσα έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινώ ευχαριστώντας τους συναδέλφους για τις πολυάριθμες τροπολογίες, 262 συνολικά που έχουν κρατηθεί. Και περισσότερες από αυτές έχουν να κάνουν περισσότερο με την προσέγγιση της έκθεσης, δηλαδή επιδιώκουν να εμπλουτίσουν το κείμενο. Ευχαριστώ τους και συγκητές για την πολύ επικοδομητική του στάση και κατά τη διατύπωση των ε, τροπολογιών μπορέσαμε χάρη σε αυτήν να προχωρήσουμε σε κείμενα τα οποία νομίζω διευκολύνουν τη δουλειά των συναδέλφων. Τώρα σε μια προκαταβολική, προκατακτική καλύτερα παρατήρηση. Πολλοί συνάδελφοι είχαν εκφράσει όταν αρχίσαμε τη μελέτη του θέματο αυτού ανησυχίε ως προς το σεβασμό τη αρχής επικουρικότητα. επικουρικότητας. Και είχαν υποβληθεί σχετικά τροπολογίε. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι το κείμενο το οποίο τώρα έχουμε πλέον ε, είναι σύμφωνο με το πνεύμα του άρθρου 195 της συνθήκης, το οποίο ξεκάθαρα ορίζει ποιες είναι οι αρμοδιότητες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ως προς την ανάπτυξη της στρατηγικής για τον ε, τουρισμό. σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας. Δεν μπορώ βέβαια τώρα να υπησέλθω στις λεπτομέρειες των 262 τροπολογιών. Θα προσπαθήσω να σας τις παρουσιάσω σε ομάδες. Κάποιες στόχο έχουν να συμπληρώσουν ε, παραδο... παραγράφους ε, προσθέτουν δηλαδή ένα κομμάτι κειμένου, διευκρινίζουν ενδεχομένω. Αυτέ θεωρώ θετικέ τροπολογίε και μπορώ να τι κάνω δεκτέ, είτε στη διατύπωση που έχουν ζητήσει οι συντάκτε του, είτε με κάποια συμβαστική τροπολογία που ενσωματώνω και πιστεύω λαμβάνει υπόψη το πνεύμα των τροπολογιών. Και μάλιστα εκεί που βλέπω ότι οι περισσότερε τροπολογίε έχουν ε, ε, το ίδιο, ε, τον ίδιο στόχο, τροπολογίες Φερρυπίν για τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Πρόβλημα γνωστό, πρόβλημα για το οποίο η Επιτροπή μας έχει ιδιαίτερη ευαισθησία επιδείξει. Άλλο η ομάδα τροπολογιών σε αυτό το, με αυτό το χαρακτήρα είναι οι τροπολογίες σχετικές με τη στρατηγική του 2020 και την αναζήτηση ενός τρόπου αλλά και συγκεκριμένων προθεσμιών για την στρατηγική για το τουρισμό που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε ήδη με διάφορες ε, δράσεις που αναπτύχθηκαν στο παρελθόν επισημάνει πως θέλουμε μια γενικότερη στρατηγική και έχουμε δώσει κάποιες ενδείξεις προς τα που θα πρέπει να βαίνει αυτή. Από την άλλη όμως υπάρχουν κάποιες τροπολογίες οι οποίες βλέπω να επιμένουν σε κάποιες ιδέες που ήδη έχουν εκφραστεί μέσα στο κείμενο ε, για αυτή την ομάδα των απολογιών θα προσπαθήσω ακόμα αυτή την εβδομάδα να έρθω σε επαφή με τους συντάκτες τους ώστε να δω εάν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμβαστική ε, πρόταση μαζί είτε εν πάση περιπτώσει να βρούμε μια λύση για την καλύτερη διατύπωση και έτσι να διευθετηθεί αυτό το θέμα ή αυτά τα θέματα που καλύπτουν αυτές τροπολογίες. Όπως και η κυρία Φώστερ ε, είδα και εγώ κάποια προβλήματα μετάφρασης στο κείμενό μου, πάλι στα αγγλικά και άρα θα πρέπει σε συνεννόηση και με τη γραμματεία να κοιτάξουμε να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα. μικροπροβλήματα τα χαρακτηρίζω. Και να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα ασάφειας ως προς την μετάφραση ορισμένες φορές στα κείμενα και αν μπορούμε με κάποια τροπολογία ε, να διευκρινίσουμε κείμενο το οποίο δεν ήταν πολύ σαφές στην αρχή. Επίσης θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε κάποιες ε, τροπολογίες, πάλι θεματικά τις παρουσιάζω, ε, όπου βλέπω να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι συνάδελφοι. Πρώτο θέμα, η τουριστική θεώρηση διαβατηρίου. Έχουμε επισημάνει διότι διαπιστώνονται δυσκολίες ως προς την χορήγηση θεώρησης τουριστικής, ε, ιδιαίτερα και κάποια αναδυόμενα κράτη προβλήματα τα οποία ενδεχομένω και να υπονομεύουν ε, την ε, ε, δυνατότητα ανάπτυξη δραστηριοτήτων των δικών μα τουριστικών επιχειρήσεων. Προτείνονται λοιπόν τροπολογίε από κάποιου συναδέλφου με διατυπώσει πιο συγκεκριμένε μερικέ φορέ στο θέμα αυτό και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε στι προσοχέ εβδομάδε να καταλήξουμε σε συμβαστικό κείμενο, δεδομένου ότι ο στόχο είναι κοινό. Συμφωνούμε στο στόχο. Επίση, Ω προ την πρόταση για αξιοποίηση κάποιων μεγάλων διεθνών εκδηλώσεων. Με στόχο την προβολή της Ευρώπης ως τουριστικού ε, προορισμού. Πάλι πιστεύω ότι μπορούμε μαζί με τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό να βρούμε συμβαστικές λύσεις. Για τη 16η όμως παράγραφο, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας επισημάνω ένα θέμα που το βρίσκω πολύ σημαντικό. Διότι όλοι θέλουμε να αποφύγουμε την υπερβολική διάδοση σημάτων, προβολής δηλαδή, ε, την, τον υπερβολικό κατακαιρματισμό τους, έτσι ώστε να έχουμε πιο συγκεντρωμένη ε, πολιτική και στρατηγική στο θέμα αυτό της προβολής μέσω ενός σήματος, μέσω ενός label. Άρα πιστεύω ότι η ιδέα για ένα ειδικό σήμα βιωσιμότητας έχει καλυφθεί κατά τρόπο στο συνθετικό στο κείμενό μου και ε, μακροπρόθεσμα νομίζω θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε τη βιωσιμότητα να την εκφράσουμε σε όρους ποιότητας. Δηλαδή όταν, όπου βλέπουμε σήμα βιωσιμότητας να ισοδυναμεί αυτό και με σήμα ποιότητας. Για να μην υπάρχουν χιλιάδες σήματα τα οποία κανείς δεν αναγνωρίζει τελικά και μπερδεύεται ο χρήστης ή ο επιχειρηματίας του τουρισμού κτλ. για το τι πρέπει να χρησιμοποιήσει, τι σημαίνει αυτό που βλέπει. Και επίσης θα ήταν καλό νομίζω, όπως είπα, να αποφύγουμε ε, αυτή την πληθώρα σημάτων για, για έναν λόγο, γιατί μερικές φορές είναι και δυσνόητα, δεν καταλαβαίνουμε τι ε, ρόλο έχουν. Για την παράγραφο 18 τώρα. Η τροπολογία 111, Σίμψον η σχετική με τις πτυχές ασφαλείας ε, στα ξενοδοχεία. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Βλέπω το στόχο που επιδιώκει ο Πρόεδρος Σίμψον με την τοπολογία αυτή. Τον ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ επίσης και τους συναδέλφους που συνέβαλαν με τις προτάσεις τους στο θέμα του ε, συσχετισμού, της υπογράμμισης του σχετισμού μεταξύ τουρισμού και μεταφορών. Είχα πει στο αρχικό μου κείμενο ότι θα πρέπει ιδιαίτερως να τονίσουμε αυτή την πτυχή Δυστυχώς όμως δεν τα καταφέραμε και έτσι βλέπω με πολύ ενδιαφέρον αυτές τις ε, προτάσεις. Και επίσης ιδιαιτέρως ως προς το θέμα των ε, ζωνών εκείνων που είναι κάπως πιο αποκλεισμένες, που δεν ευνοούνται από τις μεταφορές. Αυτές θα προσπαθήσουμε να τις ενσωματώσουμε. Ένα άλλο θέμα που δεν ήθελα να σα επισημάνω σήμερα επίση είναι ο τουρισμός για τον καθένα. Ο τουρισμός ως βιώσιμη δραστηριότητα μέσα από την ε, ιδέα του καλυψώ. Και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε ακριβώς σε αυτό κάποια θετικά ε, στοιχεία που υποστηρίζουν οι συνάδελφοι. Θέλουν δηλαδή να επεκταθεί αυτή η εμπειρία και σε άλλες ε, χώρες και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και εγώ σε αυτό θα ήμουν πιο προσεκτικός. Γιατί? Διότι βλέπω ότι το 2011 ο προπολογισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει μόνο 1,5 εκατομμύριο για την ανάπτυξη του Καλυψό το οποίο ως πρόγραμμα εκπνέει φέτος το 2011. Μεγάλο μερίδιο δηλαδή των κονδυλίων στόχο έχουν να επιτρέψουν την συνέχιση της λειτουργίας του αλλά σε μια υπόθεση περιορισμού των κονδυλίων, αφού δεν είναι σαφής ακόμη η στόχη, το να προβλέψουμε επέκταση του καλυψό ώστε να καλύψει και τρίτες χώρες, νομίζω ότι πια είναι υπερβολικό και είναι άλμα στο κενό λίγο πολύ. Και για να τελειώνω, Πρόεδρε, η ιδέα του Ευρωπαϊκού Σήματος, το Brand Europe που λέμε, η ιδέα αυτή του, της μάρκας που μπορεί να είναι η Ευρώπη, πρέπει να είναι σαφής, πρέπει να είναι ξεκάθαρη, δεν μπορεί να είναι αμφίσιμη. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο σε συγκεκριμένο μέσων ή σε συγκεκριμένο προορισμό. Πρέπει να είναι κάτι που χαρακτηρίζει, χαρακτηρίζει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αποτελεί ένα σήμα απευθυνόμενο προς τα τρίτα κράτη ή τα αναδυόμενα. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς δεν έχουμε συγκεκριμένα αναφερθεί σε ε, προορισμούς, γιατί δεν θέλουμε να προτιμήσουμε τον έναν έναντι του άλλου. Θέλουμε να προβάλλουμε την Ευρώπη ως έναν προορισμό τουριστικό, να προβάλλουμε το τουριστικό προϊόν που είναι η Ευρώπη. Και κάτι άλλο, μια σειρά τροπολογιών ως προς τα δικαιώματα των ε, τουριστών που έχω δει, ζητούν συγκεκριμένη ε, νομοθεσία για τα δικαιώματα των ε, τουριστών. Εγώ πάλι θα ήμουν εδώ επιφυλακτικός, διότι πρέπει ε, να εισαχθεί, πρόκειται να εισαχθεί ένα μέσο για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών σε κάθε είδους, ε, σε κάθε τρόπο μεταφοράς. Εδώ πάλι εδώ και καιρό ζητούμε μία προστασία των ε, επιβατών, μάλλον των ταξιδιωτών, των τουριστών σε περίπτωση πακέτου ταξιδιωτικού και αυτό πρόκειται να γίνει πολύ γρήγορα. Υποτίθεται. Τώρα το να ζητήσουμε μια ειδική νομοθεσία για το δικαίωμα του τουρίστα για τα δικαιώματα του τουρίστα. Ενώ βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα νομοθετήματα σχετικά, σημαίνει ότι ενδέχεται να ε, μην επιτύχουμε το στόχο μας όπως θα τον θέλαμε. Να υπάρξει διάχυση δηλαδή των ε, προσπαθειών μας. Αυτά, αλλά βέβαια είμαι στη διάθεση των συναδέλφων. Ο κύριος Δανέλης παρακαλώ εκ μέρους της πολιτικής του ομάδας και δεν θέλω να πω ότι έχουμε οκτώ είδη εγγεγραμμένους στον κατάλογο, γι' αυτό σας παρακαλώ σύντομα, κύριε Καδανέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, θα είμαι πολύ σύντομος γιατί ο συνάδελφος ε, Φιντάντσα αναφέρθηκε σχεδόν στο σύνολο των ε, ε, θεμάτων που μας απασχόλησαν σε αυτή την έκθεση. Θέλω να τον ευχαριστήσω για την, και την αρτιότητα και την πολύ καλή ποιότητα αυτής της έκθεσης, αλλά και την στενή συνεργασία που είχαμε σε όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας της, όπως επίσης και τον ε, συνάδελφο Ουτζίας, τον ε, ε, σκιώδη συγητή της Άλντε, για την στενή συνεργασία μεταξύ μας που φαίνεται και από τον αριθμό των κοινών τροπολογιών που έχουμε καταθέσει. θέλω να σημειώσω ότι, όπως είπα, το κείμενο είναι πλήρες και πολύ καλό ε, και γι' αυτό το λόγο η, μεγάλη πλειοψηφία των ε, πολλών τροπολογιών βελτιώνουν ή συμπληρώνουν χωρίς να αλλάξουν το νόημα, χωρίς να παρεμβαίνουν ε, αρνητικά στην έκθεση. θα σημειώσω μονάχα ότι οι περισσότερες από τις κοινέ μας τροπολογίες αφορούν σε ζητήματα της αναγκαιότητας ε, στήριξης με χρηματοδοτικά εργαλεία συγκεκριμένα των δράσεων για τον τουρισμό, τουλάχιστον για την επόμενη προγραμματική περίοδο, ε, για την αναγκαιότητα προκύπτει για την ανάπτυξη και την εξειδίκευση νέων μορφών τουρισμού, αλλά ενίσχυσης και ποιοτικής αναβάθμισης των ήδη φυσταμένων, τη δημιουργία ευνοϊκότερου συνολικά περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του τομέα, με την καινοτομία ή τις συνεργασίες των κρατών μελών, ε, καθώς επίσης ε, ένα κομβικό ζήτημα που φάνηκε από την πληθώρα των τροπολογιών είναι αυτό το οποίο ανέφερε και ο Κάρλο πριν ε, για την αναγκαιότητα της διευκόλυνσης και απλοποίησης της έκδοσης τουριστικής βίζας ε, κυρίως από τις χώρες BRIC. Τέλος, ζητούμε από την Επιτροπή να μας προδιαγράψει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των 29, των 21 ε, φιλόδοξων δράσεων για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Ε, δεν νομίζω ότι είναι ανάγκη να αναφερθώ σε άλλες επιμέρους τροπολογίες. Θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να συζητήσουμε μετά την ε, ολοκληρωμένη εργασία που έχουμε. Ε, όμως να σημειώσω ότι ε, συνάδελφοι από όλες τις πολιτικές ομάδες έχουν καταθέσει πολύ ενδιαφέρουσες ε, τροπολογίες. Ευχαριστώ. Thank you for the Mr. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας τον Κάρλο Φιντάντσα. για ένα πολύ καλό κείμενο. Τον συγχαίρω για τη μέθοδο που ακολούθησε. δεν πρέπει να τον εκπλήσει ο αριθμός των τροπολογιών. Είναι σημείο ότι ο κόσμος δίνει προσοχή στο θέμα αυτό. Είναι ένα καινούριο θέμα. Είναι πρώτη φορά που ασχολούμαστε με αυτό, γιατί μόλις τώρα έχει ενταχθεί στην συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Και όπως και ο Σπύρος Δανέλης, θα ήθελα και εγώ να πω ότι όλοι οι σκιώδεις ε, οι συμφώνησαν και αυτό είναι γιατί είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξαρτιέται όλο ένα και πιο πολύ από την ανάπτυξη της οικονομίας μέσα από τον τουρισμό με θετικό τρόπο. Και πιστεύω ότι αν ακολουθήσουμε αυτό που κάνουμε σε αυτή την έκθεση θα είμαστε σε θέση να σαγάγουμε το ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό σύστημα, κάτι το οποίο χάσαμε τους τελευταίους αιώνες ως αποτέλεσμα ανάπτυξης σε άλλες υπήρους. Νομίζω ο τουρισμός είναι ένα περίπλοκο θέμα. Δεν το συνειδητοποιούμε πάντα πόσο περίπλοκο θέμα είναι, αλλά θα το δούμε και στο μέλλον καθώς αναπτύσσουμε την κοινοβουλευτική μας δράση σε αυτό τον τομέα μελλοντικά. Ωστόσο, η έκθεση και οι τροπολογίες δείχνουν ότι έχουμε παρομοίες προσεγγίσεις μακροχρόνια είναι μια στρατηγική στην οποία θα ενταχθούν όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υποδείξω ότι σε σύγκριση με το αρχικό κείμενο βλέπουμε βελτιώσεις. Για παράδειγμα, η εισαγωγή της ιδέας ότι ο τουρισμός είναι ένα σύστημα. Είναι ένας ε, ολοκληρωμένος μηχανισμός όπου συμμετέχουν άλλοι παραδοσιακοί τομείς. Και αυτό είναι το δυνατό σημείο αυτού του κειμένου. Ναι, οι παραδοσιακοί τομείς θα δραστηριοποιηθούν μέσω του τουρισμού. Και πάλι, εντάξει. θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εισαγαγεί μια ε, σφαιρική στρατηγική τουρισμού μέχρι το 2012. Μιλούσαμε για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Πιστεύω ότι θέλουμε και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα του τουρισμού. Ο τουρισμός είναι εποχιακός σε πολλές περιφέρειες της επικράτειας της Ευρώπης. Θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική για να το υπερπηδήσουμε αυτό το ε, πρόβλημα και να έχουμε και μια πολιτική που να ενσωματώνει παροδοσιακές τουριστικές περιοχές με άλλες περιοχές, πλούσιες και φτωχές περιοχές. Θα κλείσω εδώ και όταν μιλήσουμε στις τροπολογίες, για τις τροπολογίες θα πάρω το λόγο. Σας ευχαριστώ για τους περάσινους, κυρία Πρέπολς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και νομίζω ότι ο αριθμός των τροπολογιών που επευλήθησαν στην έκθεση του κυρίου Φιντάντσα αποτελεί απόδειξη πως ο τουρισμός είναι τομέα σημαντικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε τώρα πιστεύω αντιμέτωποι με μια μεγάλη πρόκληση, χάρη δηλαδή σε αυτές τις ε, τροπολογίες να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ε, προτεραιότητα σε μια ε, έκθεση γνώμη, όπου να προσδιορίζονται οι προτεραιότητε για τον τουρισμό με βάση βέβαια και τους όρους της ε, συνθήκης του άρθρου 195 συγκεκριμένα. Και θα ήθελα εκ μέρους των ε, Πρασίνων να εκφράσω τη διάθεσή μας, τη θεσιμότητα μας καλύτερα να συνεργαστούμε με τον εισηγητή στην διατύπωση συμβαστικών τροπολογιών. Έχει άλλωστε και ο ίδιος πει ότι συνεχίζει αυτή την προσπάθεια και τη συζήτηση. Κάποια σημεία τα οποία βρίσκω ενδιαφέροντα και είναι σημαντικά για την ομάδα μας και τα συναντώ και σε τροπολογίες άλλων συναδέλφων είναι τα εξή. Καταρχάς ποιότητα και ε, διάρκεια. Πριν από μερικές εβδομάδες εδώ στο Κοινοβούλιο είχαμε ένα συνέδριο που οργάνωσα εγώ για τον τουρισμό. Ως φλαμανδί λοιπόν προσπάθησα να προβάλλω κάποιες πρακτικές και η παρουσίαση απέδειξε ότι η ποιότητα και η διάρκεια στον τομέα του τουρισμού μόνο θετική μπορεί να αποβεί για κάθε έναν εμπλεκόμενο. Άλλωστε όλοι οι εκπρόσωποι που είδαμε και από άλλες περιοχές ακόμη ε, μας έκαναν θετικά σχόλια και για την πρόσβαση και για την ποιότητα και για τη διάρκεια. Άρα αυτό ενισχύει την ε, πεποίθησή μου ότι θα πρέπει αυτά τα στοιχεία να είναι χαρακτηριστικά τη όποια πολιτική για τον τουρισμό να αναπτύξουμε στο μέλλον. Αυτή είναι η προσθέμενη αξία στη τελευταία ανάλυση που μπορούμε να δώσουμε εμεί. Και για το κριτήριο ποιότητα. θα ήθελα να υπογραμμίσω τι τροπολογίε υπαριθμών 7 και 224. Για δε την διάρκεια, οι 157 και 158 τροπολογίες μου φαίνονται πολύ σημαντικές και θα παρακαλέσω επίσης να γίνεται καλύτερο τονισμό μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων που άλλωστε σαφώς ζητάει το άρθρο 195 της συνθήκης. Αυτό λέω και στι μου. Επίσης και ο κύριος Φιντάντσα το υπογράμμισε ήδη. Η έκθεση θα πρέπει να αποτελεί μια επικοδομητική λύση να προσφέρει μια επικοδομητική λύση ως προς το θέμα της μάρκας του σήματος μια επικοδομητική λύση λοιπόν, μια αποτελεσματική πρόταση χρειάζεται, όπως άλλωστε είχα πει και την προηγούμενη φορά, ε, Φερρυπίν με την θέσπιση του χάρτη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του τουρίστα που είχαν ε, κάνει δεκτή ως ιδέα και οι συνάδελφοι και η Επιτροπή. Αυτά τα επαναφέρω στην σχετική τροπολογία, διότι πιστεύω ότι, πάρει, είναι διαφορετικό το θέμα των δικαιωμάτων του τουρίστα και εκείνο των επιβατών που θα πρέπει να υπογραμμιστούν. Ευχαριστώ κύριε Φώστη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φιντάντσα, τον εισηγητή. Είναι προφανώς, είναι τεράστιος ο αριθμός των τροπολογιών όπως είπατε και χρειάζεται να καταβάλουμε προσπάθειες για να καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στους κέριους τομείς που διαλαμβάνει αυτή η έκθεση. Αλλά προφανώς ο κ. Φιντάντσα προσπαθεί να το κάνει αυτό. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα σημεία τα οποία ήθελα να θίξω. Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε εδώ πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός για τα περισσότερα από τα κράτη-μέλη μας, για όλα τα κράτη-μέλη μας. Και είναι πολύπλοκο το πρόβλημα του τουρισμού γιατί εμπλέκει πάρα πολλές πτυχές, είτε είναι οι μεταφορές, είτε είναι τα ξενοδοχεία κτλ. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί για το πώς θα προχωρήσουμε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παραδείγματος χάρη, στο Ηνωμένο Βασίλειο <clears throat> ο τουρισμός είναι μια αποκεντρωμένη αρμοδιότητα της Σκοτίας, της Αγγλίας, της Ιρλανδίας κτλ. Επομένως, δεν θα υπάρξει θετικό πνεύμα για να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις λεπτομέρειες και τη μικροδιαχείριση του τουρισμού σε τοπικό επίπεδο. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Επίσης, εμείς χαιρετίζουμε τη βασική αυτή κατευθυντήρια γραμμή της έκθεσης και κάποιες από τις τροπολογίες της. Τονίζω όμως και πάλι <clears throat> με τόσες τροπολογίες πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην έχουμε τροπολογίες οι οποίες ουσιαστικά λένε ελάτε στη χώρα μας, ελάτε στην τάδε περιοχή, ελάτε στο τάδε χωριό κτλ. Αυτό συμβαίνει βέβαια πολλές φορές με τις τροπολογίες αυτό το οποίο είναι σημαντικό εξάλλου, να εξασφαλίσουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες εμπλέκονται στον τομέα του τουρισμού και είναι πολλές και πιστεύουν ότι έχουν τεράστιο άχθος ρύθμισης, να προσπαθήσουμε να, τους, να τις βοηθήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη των οικονομιών μας. Να μην επιβάλλουμε λοιπόν πρόσθετο βάρος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, η Κομισιόν θα πρέπει να εστιάσει σε προτεραιότητες οι οποίες προωθούν την καινοτομία και μειώνουν το άχθος πάνω στις επιχειρήσεις. Θα ήταν χρήσιμο η Κομισιόν επίσης να μας δώσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έχουμε το σχέδιο με 21-22 σημεία, αλλά να μας πει ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας για την υλοποίηση αυτών των στόχων να έχουμε μια καλύτερη εικόνα λοιπόν για όλα αυτά. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί επίσης και με τις ετικέτες, <clears throat> με τα σήματα. Έχουμε διαδικασίες για την απονομή σημάτων στα κράτη-μέλη και ίσως θα ήταν θετικό να έχουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να το κάνουμε όμως αυτό με προσεκτικό τρόπο και δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια πολυπικιλία και πληθώρα σημάτων, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε σύγχυση και για τους επαγγελματίες, αλλά κυρίως για τον καταναλωτή. Ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο όταν μιλάμε για ε, εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα αυτό, θα πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι μετακινούνται από ένα κράτο σε άλλο για να αποκτήσουν εμπειρία στη δουλειά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα τελικό σημείο υπάρχουν θέματα τα οποία δεν αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον τουρισμό, όπως είναι το θέμα της, ε, των προξενικών θεωρήσεων, έχει να κάνει και με εθνική ασφάλεια και με άλλα προβλήματα. Ίσως όμως θα μπορούσαν τα κατημέλη να βελτιώσουν αυτές τις διαδικασίες μόνα τους, όχι να μπει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα και να λέει στα κράτη-μέλη τι πρέπει να κάνουν. Σίγουρα θα μπορούσε να υπάρχει μια μεγαλύτερη ευκαμψία για τα θέματα αυτά. Και για την οδηγία για τις διακοπές πακέτο, για τα ταξιδιωτικά πακέτα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Και τέλος για την καλυψό και τον κοινωνικό τουρισμό. Εάν τα κράτη-μέλη θέλουν να έχουν τα δικά τους προγράμματα, εάν θέλουν να δαπανίσουν εθνικά κονδύλια για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που πηγαίνουν διακοπές, αυτό είναι δικό τους θέμα. Στο πρόγραμμα Καλύψο έχουν δοθεί 100, 1 εκατομμύριο ευρώ <clears throat> το 2009 για το πρόγραμμα αυτό. Θα ήθελα να ξέρω όμως ποια ήταν η κατανομή αυτών των κονδυλίων. Θα ήθελα να τα ξέρω αυτά, γιατί <clears throat> το ερώτημα είναι αν πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις διακοπές των πολιτών. Δεν ξέρω αν αυτό είναι η δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν άλλη άποψη, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό είναι στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εγώ πάντως θέλω να υποστηρίξω τον εισηγητή, κάνει πολύ καλή δουλειά και θέλω να τον ευχαριστήσω και αυτόν και εσάς για την ε, έκθεση <clears throat> που έφερα και για την υποστήριξή σας στην έκθεση που έφερα εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον τουρισμό. Ευχαριστώ πολύ. Uh, σας ευχαριστώ κύριος Δεγράνδες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα και στο παρελθόν να επενέσω τον κύριο Φιντάνσα για την έκθεσή του, αυτό με την ευκαιρία της πρώτης συζήτησης που κάναμε για το θέμα αυτό. τουρισμός είναι πολύ σημαντικός για τις χώρες μας και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό γιατί ο τουρισμός είναι όχι μόνο μία πηγή εσόδων για τις οικονομίες μας που πλήττονται από την οικονομική κρίση, αλλά κύριε Πρόεδρε είναι και ο καλύτερος τρόπος για να πλησιάσουν ο ένας τον άλλο οι πολιτισμοί και να υπάρχει καλύτερη κατανόηση των λαών. Γι' αυτό οι τροπολογίες που έχουμε ε, παρουσιάσει ε, στην έκθεση αυτή έχουν αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλουν λοιπόν να τροποποιήσουν την γραμμή του κ. Φιντάνσα, αλλά να προσθέσουν ορισμένε ιδέε που δείχνουν τι δυνατότητε που έχουμε στην Ευρώπη και ιδίω μετά από την έγκριση τη συνθήκη τη Λισαβόνα να υπάρξει και μια συμπλήρωση των εθνικών πολιτικών στον τομέα του τουρισμού. Πρέπει να δούμε για τις ε, βοήθειες που δίνονται σε κρατικό επίπεδο, αν μπορούμε να τις ε, καταργήσουμε όλες ή αν πρέπει να τις διαμορφώσουμε και όλα αυτά. Υπάρχουν θέματα όπως ο κοινωνικός τουρισμός, η εδαφική συνοχή, οι περιοχές που έχουν την ε, σωστή, <clears throat> έχουν ε, συγκριτικό πλεονέκτημα και επίσης τα θέματα της υποστήριξης με την, ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συνάδελφό μου η Ρώσα Στεργά που έρχεται και από την περιοχή των Βαλεαρίδων που είναι μια από τις πιο τουριστικές περιοχές στον κόσμο μπορεί να σας πει περισσότερα λεπτομεριακά για τις τροπολογίες αυτές, που νομίζω ότι βοηθούν ιδιαίτερα να προωθήσουμε τον τουρισμό στην Ευρώπη. Κάτι πολύ σημαντικό. Θέλω λοιπόν και πάλι να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη θαυμάσια εργασία του και το στόχο να γίνει η Ευρώπη ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο. Αυτό είναι φιλόδοξο, αλλά εφικτό και η έκθεση αυτή πρέπει να βοηθήσει να επιτύχουμε το στόχο αυτό. Ευχαριστώ. Κυρία Μάισνερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά του. Έχουμε δύο νέε αρμοδιότητε δυνάμει τη συνθήκη Λισαβόνα Και βέβαια ακούγεται το ερώτημα πάντα γιατί αφού υπάρχει ο τουρισμό στην Ευρώπη ήδη και μπορεί να τον ρυθμίσουν τα κράτη-μέλη, γιατί να χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό τουρισμό. Το ακούμε πολλέ φορέ και στη Γερμανία. Κοιτάξτε να σα πω, πρέπει να βρούμε ακριβώς αυτό το σημείο στο οποίο μπορούμε να δώσουμε κάτι περισσότερο στην Ευρώπη για εκείνον τον οποίο, ο δεν έχει τόσο πολλά ε, τόσο μεγάλη οικονομική επιφάνεια, ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό ε, βιοπορισμό, ένα σημαντικό οικονομικό παράγοντα και αυτό νομίζω θα πρέπει ακριβώς να κοιτάξουμε ως πτυχή που μπορεί να προβάλλει η Ευρώπη ως ε, τόπος δηλαδή ως προορισμός τουριστικός η Ευρώπη μπορεί να κοιτάξει και αυτή την πτυχή. Έχουμε μεγάλο τουρισμό. Κάποιοι λένε ναι γιατί να κάνουμε κάτι περισσότερο χρειαζόμαστε περισσότερους τουρίστες. Βεβαίως το πρέπει να το δούμε όμως αυτό και να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες και να διαπιστώσουμε, να εντοπίσουμε τι το διαφορετικό έχει να, προσθέσει, να προσφέρει η Ευρώπη, τι τους διαφορετικό τουρισμό μπορούμε να δούμε, να αναπτύξουμε φερρυπίν βιομηχανική κληρονομιά που ανέφερε ο συνάδελφος ο πρόεδρος, άλλες ιδέες που θα πρέπει να κοιτάξουμε και την ιδέα του σήματος, του label που θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε περαιτέρω τι μπορούμε να δαχθούμε ένα από τον άλλον, ε, χωρί βέβαια επιπλέον γραφειοκρατία του αντίο, να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία και εδώ έχει δίκιο η κυρία Φώστερ, για να στηρίξουμε ακριβώ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει που απασχολούν στο τομέα αυτό, να μπορούν να βρουν μια θέση στον ήλιο. Και ε, σαν σήμα. Να σας πω, υπάρχει φερειπίν σε όλο τον κόσμο η ιδέα του romantic hotel, του ε, παλιού εκείνου σπιτιού που είχε ωραία διακόσμηση κτλ. ή του αντίστοιχου castle στην ε, Αγγλία, παλιά κάστρα που έχουν τραπήσει ξενοδοχεία, του παραδόρ στην Ισπανία. αυτά όλα λοιπόν μπορούμε νομίζω να τα δούμε σαν κατηγορίες τουριστικές τις οποίες μπορούμε να στηρίξουμε το ευρωπαϊκό σήμα. Και θέλουμε μία ε, ιδέα του τουρισμού στην Ευρώπη, η οποία είναι ελκυστική και για τον Ευρωπαίο, αλλά και για εκείνον που έρθει από τον υπόλοιπο κόσμο και θα παρουσιάζει ε, την Ευρώπη κατά τρόπο ελκυστικό. Ο κύριος Μπάχ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι ιδιαίτερος δεν θέλω να εκφράσω τις ευχαριστήσεις μου στον κύριο Φιντάντσα για την έκθεσή του. Είναι σαφές ότι κατέχει το ζήτημα πολύ καλά και μάλιστα με πολύ πάθος ε, το πραγματεύεται. Οι πολλές τροπολογίες νομίζω ότι αποτελούν απτή απόδειξη και μόνο αυτού, ότι δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον τουρισμό. Πολλά ε, υπόθηκαν ήδη, θα επικεντρωθώ μόνο σε αυτά που με ενδιαφέρουν περισσότερο. Δεν πρέπει να λησμονήσουμε την ιδέα που εκφράζεται και με τις εθνικές θέσεις τις εθνικές εκδηλώσεις ότι ε, πρέπει να τις τονίσουμε αυτές τις ιδέες, αυτές τις δραστηριότητες μέσα από ένα ευρωπαϊκό ε, πνεύμα. Επίσης, ο τουρισμός με δεδομένες δημογραφικές εξελίξεις ανά τον κόσμο θα πρέπει να υποστηριχθεί για διάφορους λόγους και σε, διάφορους, σε διάφορες κατηγορίες τουριστικές, φερρυπίν ιατρικό τουρισμό, με ρυθμίσεις που θα πρέπει να λάβουν φυσικά να διπεραιώσουν με ρυθμίσεις τους οι άλλες ε, επιτροπές του Κοινοβουλίου, ε, φερρυπίν για ανάληψη των, ε, του κόστους των δαπανών των ιατροφαρμακευτικών, ε, αναγνώριση ασφάλισης ιατροφαρμακευτικής ε, ένθρακα και τα συνόρων κτλ. Αυτό λοιπόν είναι, είναι μορφές του τουρισμού που θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Ένα άλλο ζήτημα που θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης και έχει να κάνει με τις Αρδένες, γιατί δεν έγραφα για τις Αρδένες ε, την τελευταία εβδομάδα. Ε, είναι μια περιοχή, Φερρυπίνη Αρδένες, οι οποίες ανήκουν σε τρία-τέσσερα διαφορετικά κράτη. Ε, αυτές, σαν πρότυπο για τον ευρωπαϊκό τουρισμό, νομίζω μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ καλό παράδειγμα. Και θα πρέπει να το εξετάσουμε περισσότερο τι έχει γίνει εκεί. Ιδιαίτερα επίσης καλή μου φαίνεται η ιδέα της ε, κατάρτισης ή της ε, επιμόρφωσης για τους εργαζομένους στον τουρισμό ώστε να βελτιώσουν τη δυνατότητα να υποδεχθούν τον ε, τουρίστη. Ευχαριστώ. κυρία Σεχμάλοβα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ επί τη ευκαιρία να συγχαρώ τον εισηγητή μας. Η δουλειά του είναι πολύ καλή και είναι δουλειά σε ένα νέο τομέα, περίπλοκο. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με την Ευρώπη που θέλουμε να καταστήσουμε τουριστικό πρόεδρο υπαριθμών ένα για ολόκληρο τον κόσμο, ήδη είναι στην πρωτοκαθεδρία και θα ήθελα ιδιαίτερος να υπογραμμίσω την ανάγκη για μια πιο απλή πολιτική για τη θεώρηση διαβατηρίου, για πιο εύκολη χορήγηση της θεώρησης, αλλά και για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφορών περιφερειών, διότι οι περιφέρειες θα πρέπει να μην είναι μόνο ανταγωνιστικέ μεταξύ τους, μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους και αυτό είναι προς του τουρισμού. Καλή ιδέα επίσης βρίσκω το να κοιτάξουμε να βρούμε νέες ομάδες στόχους. Φερρυπίν, κοινωνικός τουρισμός, τουρισμός ατόμων με αναπηρίες και ούτω καθεξής. Είναι ιδέες που θα πρέπει να διερευνήσουμε. Θα συμφωνήσω εδώ με την κυρία Φώστερ ως προς το ότι χρειάζεται να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να εξασφαλιστεί αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε όλη την Ευρώπη, αμοιβαία δηλαδή. Πολλές φορές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τον πρώτο ε, εργοδότη που θα προσλάβει κάποιο νεαρό ή κάποια γυναίκα σε μια τέτοια δουλειά. Κύριο Κράμερ, ευχαριστώ. Για την τροπολογία 272 θα ήθελα να λάβω το λόγο ζητώντα συγγνώμη γιατί δεν την έχω συντάξει εγώ. Είναι μια πολύ καλή πρόταση που ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει στη δικτύωση και συνεργασία μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αναπτυχθούν τα περιφερειακά εκείνα συμβούλια που θα ενισχύσουν την ε, οικολογική διάσταση του τουρισμού στην Ευρώπη. Δεν είναι δική μου όπως τροπολογία, αλλά είναι πάρα πολύ καλή στην πραγματικότητα. Ω, έτσι δεν είναι. Όχι, πείτε μου κυρία Μάισνερ, δεν είναι πολύ καλή. Είναι πολύ εύστοχα όλα αυτά. Έχουμε πολύ καλά συμβούλια λοιπόν, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να έχουμε πολύ καλά δίκτυα ποδηλατικά, ποδηλατοδρόμων δηλαδή, που μπορούμε να προβάλλουμε και για τον τουρισμό, για ε, για μην ξεχάσουμε ότι μέσα από τις περιοχές αυτές είναι η μόνη τους ευκαιρία ε, το ποδήλατο, ο ποδηλάτης καλύτερα για να γνωρίσουν τουρίστες, για να δουν τουρίστες. Αυτά λοιπόν. Θέλω να επισημάνω επίση ότι εμεί ω Ευρωβουλευτέ θα πρέπει να ασχολούμαστε όχι μόνο με την εθνική, την περιφερειακή, αλλά την ευρωπαϊκή διάσταση πάνω απ' όλα και κοιτάω εδώ το Ματιού ιδιαίτερος. ιδιαίτερο. Η 72α λοιπόν είναι πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε στας Η κυρία Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ καταρχήν τον κύριο Φιντάντσα για την έκθεση αυτή που έχει εκπονήσει. Όλα αυτά τα οποία έχει αντιμετωπίσει είναι πραγματικά ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέματα και καλύπτει όλο το φάσμα των θεμάτων αυτών. Όπως είπε ο Λουίς Δεγκράντες, έχουμε καταθέσει μια σειρά από τροπολογίες, κυρίως για να τον βοηθήσουμε να συμπληρώσει την έκθεση αυτή. Και μία από τις τροπολογίες αυτές συγκεκριμένα μιλάει για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος στον τομέα του τουρισμού, κυρίως για να προωθήσουμε το επιχειρήν στον τουρισμό και επίσης τονίζουμε την ανάγκη να βελτιωθεί η χρηματοδότηση και η πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις των ε, αυτονόμων εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης τονίζουμε τη σημασία της ε, κατάρτισης και της καινοτομίας για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τη διαβίου κατάρτιση και επίση, σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο τονίζουμε την ανάγκη να ξεπεραστούν οι φραγμοί που παραμένουν ακόμα στην εσωτερική αγορά τη Ευρώπη για την πλήρη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπόριου. Σε ό,τι αφορά τα σήματα, <clears throat> η θέση του κυρίου Φιντάνσα είναι απόλυτα η ορθή, ιδίω για το ευρωπαϊκό σήμα τουρισμού ποιότητα, που έχει ένα συμπληρωματικό χαρακτήρα με τα εθνικά σήματα και δίδεται και μπορεί να το αποκτήσει κανείς με εθελοντικό τρόπο και καταθέτουμε μια τροπολογία για να υπάρξει και μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για τη σημασία των σημάτων και να μην υπάρξει υπερπληθώρα σημάτων. Μια πολύ σημαντική επίσης πρόταση του εισηγητή είναι η σταδιακή εναρμόνιση όλων των προγραμμάτων ε, πιστοποίησης και προτύπων για, την, ε, για τα καταλήματα, τα τουριστικά κτλ. Αυτό μπορεί να γίνει με την συμμετοχή του τουριστικού τομέα γιατί είναι απαραίτητο να έχουμε, μια, να έχουμε ενιαία πρότυπα σε όλη την Ευρώπη και επίσης το να αντιμετωπίσουμε την εκτός εποχής, ε, τον εκτός εποχής τουρισμό, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Ευρώπη και έχουμε καταθέσει προτάσεις για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτή τη διαδικασία και επίσης άλλες τροπολογίες όπως είπε ο κ. Δεγράντες αφορούν τις ε, νήσους ε, Βαλεαρίδες γιατί μέσα στα πλαίσια μιας πολιτικής καλύτερης σύνδεσης με τα νησιά, τα οποία είναι υπερπεριφερικά ή γενικά τα νησιά και ιδίω αυτά που έχουν μεγάλες δυσκολίες πρόσβασης, πρέπει να τονίσουμε τη σημασία των καλύτερων συνδέσεων. Και έχουμε τονίσει ακόμα το να υπάρξει μια στρατηγική όχι μόνο για τις παράκτιες περιοχές και τον παράκτιο τουρισμού, αλλά και για τα νησιά εν γέννη, γιατί στο μεγαλύτερο μέρος της τα νησιά ζουν από τον τουρισμό. <clears throat> και κλείνω λέγοντα ότι όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν τα διαρθρωτικά ταμεία καλύπτονται από τροπολογία μα, που λέει ότι στου κανονισμού εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η αναδιάρθρωση και η μετατροπή περιοχών που ήταν παλιοί τουριστικοί προορισμοί και τώρα έχουν ξεπεραστεί και πρέπει να προσαρμοστούν και να προσανατολιστούν σε νέες διαδικασίες. Ο κύριος Τέιλορ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πέντε τροπολογίες έχω καταθέσει. Αυτή που αφορούσε την κινητικότητα και την καλύτερη πρόσβαση, αυτή που αφορεί την, ε, τις προστατευόμενες περιοχές και επίσης για τους ε, συνταξιούχους να μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη πρόσβαση στα θέματα αυτά. Και επίσης είναι σημαντικός και τομέας των ζωολογικών κήπων Έχουμε περίπου 500 ζωολογικούς κήπους στα κράτη-μέλη, αλλά υπάρχουν και ζωολογικοί κήποι οι οποίοι δεν υπόκεινται σε ρύθμιση και είναι άναρχοι κατά κάποιο τρόπο. Αυτό δημιουργεί προβλήματα και για τη δημόσια υγεία και για την ευζοία των ζώων. Και χαίρομαι ότι ο Βρετανικός φορέας των ε, ταξιδιωτικών πρακτόρων αναγνωρίζει τη σημασία της ευζοίας των ζώων και έχει αναπτύξει ένα κώδικα συμπεριφοράς που ζητούμε η Κομισιό να το λάβει υπόψη. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο επανέρχεται συνέχεια στο, στη συζήτηση που είναι οι πόροι οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για τον τουρισμό. Άκουσα αυτά που είπε η κυρία Φώστα για την υποστήριξη της Βρετανικής κυβέρνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι κάπως παράξενο γιατί έχει περικόψει τον τουρισμό του περιφερειακού μου, του γραφείου της περιοχής μου, κατά του τουριστικού γραφείου της περιοχής μου, κατά 25%. Και η τροπολογία μου 245 ζητά από την Κομισιόν να αναπτύξει σαφείς κατευθύνσεις για χρηματοοικονομική υποστήριξη περιοχών που θέλουν να αναπτύξουν ε, προγράμματα τουρισμού. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν στην διαδραστική επιφάνεια του τουρισμού. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και είναι απαραίτητη η χρηματοδότηση για να μπορέσουν να αναπτύξουν περισσότερο τις τουριστικές δραστηριότητες εκεί. Πριν δώσω το λόγο στην Κομισιόν, ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Φιντάντσα για την ε, πολύ καλή έκθεσή του και ιδίως για την υποστήριξή σας στην τροπολογία 111 που αφορά την πύρα και την ασφάλεια από διοξίδιο του, από μονοξίδιο μάλλον του άνθρακα θα θυμόσαστε την τραγωδία που είχε γίνει <clears throat> με μια οικογένεια από το Ηνωμένο Βασίλειο που ένα παιδί τους δηλητηριάστηκε από μονοξίδιο του άνθρακος και γι' αυτό χαίρομαι για την υποστήριξή σας και όπως είπε και η κυρία Μάσινα, μια έκθεση τουρισμού δεν μπορεί να είναι έκθεση τουρισμού εάν δεν αναφέρεται και στην βιομηχανική μας κληρονομιά και αυτό αναφέρεται στην τροπολογία 170. Γιατί, Γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τους τουριστικούς προορισμούς. Στο παρελθόν θεωρούσαμε ότι ο τουρισμός είναι μονάχα ή οι Άλπεις ή οι παραλίες της Ευρώπης. Αλλά υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που έχει να δώσει η Ευρώπη ως πολιτιστική κληρονομιά και η πολιτιστική κληρονομιά της βιομηχανικής επανάστασης είναι ένα από αυτά τα σημαντικά στοιχεία. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν και πάλι τον κύριο Φιντάντζα και είμαι σίγουρος ότι θα περάσατε ένα θαυμάσιο Πάσχα εξετάζοντας τις 262 τροπολογίες και τώρα ο Μάικλ Λίπο θα καταθέσει μερικές ακόμα τροπολογίες για να σας βοηθήσει. Η ο κύριος έχει το λόγο. και εγώ θα ήθελα να <clears throat> χαιρετήσω την ε, μορφή που έχει λάβει πια η έκθεση του κύριου Φιντάνσα Δίνει υποστήριξη στις προτάσεις της Κομισιόν και θέτει και μερικές νέες προτάσεις μέσω των τροπολογιών των βουλευτών. Νέες προτάσεις λοιπόν και φυσικά εμείς θα δώσουμε και μεγάλη σημασία σε αυτά τα οποία ζητήσατε εσείς, δηλαδή να ε, εστιάσουμε την προσοχή μας σε ορισμένε προτεραιότητες. Σίγουρα εμείς σεβόμαστε αυτό το οποίο αναφέρετε εσείς ότι πρέπει βάσει τη συνδίκη Λισαβόνας να υπάρξει πλήρης σεβασμός της ε, επικου, <clears throat> αλλά να υπάρξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια προσπάθεια για την ε, καλύτερη εναρμόνιση και συντονισμό των εθνικών πολιτικών που να έχει και προσθέμενη αξία. Ξέρουμε πόσο σημαντικός ο τουρισμός και πώς επηρεάζει άλλες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες οικονομικές δραστηριότητες στην Ευρώπη. Και συμμεζόμαστε τις απόψεις που εκφράσαν πολλοί από εσά για την ανάγκη να διατηρήσουμε και την ποιότητα και την αηφορία γιατί είναι δύο δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και μας οδηγούν σε μια κατάσταση win-win που είναι θετικού και όχι μηδενικού αθροίσματος. Εμείς δεν μπορούμε φυσικά να παρέμβουμε συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένο επίπεδο στον τουρισμό, αυτό μας, δεν μας το επιτρέπει η συνήθεια της και δεν θέλουμε να υπάρξει υπερβολική ρύθμιση σε άλλες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς προσπαθούμε να προωθήσουμε την καινοτομία με καλύτερη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και ε, <clears throat> επικοινωνίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θέλουμε να είμαστε σε επαφή με τους επαγγελματίες του τουριστικού τομέα, με τους καταναλωτές και τα κρατη τα οποία προσπαθούν να δημιουργήσουν σήματα ποιότητας με στόχο να μην υπάρχει επικάλυψη και να υπάρχει μια γενική εθελοντική ε, παροχή ευρωπαϊκών σημάτων για το καλύψω. Εμείς προωθούμε <clears throat> τις ε, ανταλλαγές τουρισμών εκτός σεζόν για τους τουρίστες αυτούς που θέλουν να συμμετάσχουν σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Εμείς δεν έχουμε χρηματοδοτήσει άμεσα αυτές τις ε, ανταλλαγές, απλώς έχουμε εντοπίσει πρωτοβουλίες στις τέσσερις ομάδες ε, στόχου που περιλάμβανε η προπαρασκευαστική δράση και βοηθούμε να φέρουμε σε επαφή κράτη-μέλη από το Βορρά, το Νότο, Ανατολή και Δύση να ανταλλάξουν πληροφορίες, να μεταλαμβαδεύσουν πρακτικές και να προωθήσουν τις ανταλλαγές τουριστών εκτός τουριστικής σεζόν, εκτός υψηλής σεζόν. Θέλω λοιπόν να κλείσω με αυτό που είπατε <clears throat> για την βιομηχανική ε, παράδοση είναι ένα σημαντικό στοιχείο λοιπόν να διαφοροποιήσουμε τις τουριστικές μας προσφορές και εφέτος ένας από τους κύριους ε, προορισμούς θα περιστρέφεται γύρω από τα θέματα της βιομηχανικής κληρονομίας και θα είναι και αντικείμενο ενός συμποσίου που θα κάνουμε το Σεπτέμβριο. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω και εσά και τον εισηγητή και είμαι στη διάθεσή σα αν θέλετε περαιτέρω διευκρινήσει για τι πρωτοβουλίε τη Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ο Κάρλο θέλει να απαντήσει εν συντομία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και αν αφήσω κάτι πίσω τώρα θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω με τους αντίστοιχους συναδέλφους που υπέβαλαν τις τροπολογίες στη συνέχεια μεταγενέστερα και θα προσπαθήσω να εισηγηθώ συμβιβαστικές λύσεις. Στο θέμα της ποιότητας και αηφορίας, η κυρία Μπρέιπολς ανέφερε κάποιες τροπολογίες και έγινε μια σημαντική αναφορά σε περισσότερη ομοιομορφία στις διαδικασίες προειδοποίησης. Προειδοποίηση νομίζω είναι σωστός ο όρος, προειδοποίηση, warnings στα αγγλικά. Σε κάποιες χώρες όταν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, σύγκρουση, φυσική καταστροφή, η Ευρώπη κινείται σε διαφορετικές ε, ταχύτητες, οι διάφορες ε, αρχές ε, προβαίνουν σε διαφορετικές ενέργειες. Η κάθε χώρα έχει ένα διαφορετικό σύστημα προειδοποίησης. Ίσως να ήταν χρήσιμο να έχουμε μια κοινή προσέγγιση σε αυτό το τομέα. Στο θέμα των δικαιωμάτων των τουριστών θα πρέπει να επανέλθω, διότι είναι κάτι το οποίο έχει εγερθεί εκ νέου. μπορούμε να βρούμε εργαλεία τα οποία είναι ορατά και παρέχουν όσο τη δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σε τουρίστες για ήδη υφιστάμενα δικαιώματα. Ένας τουρίστας σε κάποιο το ταξίδι έχει κάποια δικαιώματα. Άλλο ο οποίο αγοράζει ε, ένα εισιτήριο σε κρουαζιερόπλιο έχει άλλα δικαιώματα. Είναι διαφορετικό συμβόλαιο αυτό και θα πρέπει να ε, ε, πληροφορούμε τους τουριστέ για τα δικαιώματά τους, τα εκάστοτε δικαιώματά τους. Τώρα, για θα μιλήσω με συναδέλφους και θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια διατύπωση και θα αποφασίσουμε ποια τροπολογία θα πρέπει να αποσυρθεί. Μιλήσαμε για παρόμοια προσέγγιση με την έκθεση του κυρίου Κουμουτσάκου. Όταν μιλάμε για το σήμα, αυτό που είπε η Κομισιόν επαρκεί. Εμείς στο κείμενο προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να προωθήσουμε ένα σύστημα διαπίστευσης, εθελούσιας διαπίστευσης από τα μέλη, το opt-in που να χρησιμοποιεί ε, το ίδιο σήμα, ένα γράμμα Q από τη λέξη quality, ποιότητα στα αγγλικά, η ιδέα είναι να προωθείτε κάτι ανάλογο και σε άλλα κράτη-μέλη για να ακολουθούνται τα ίδια ε, κριτήρια. Αλλά είναι ένα εθελοντικό σύστημα και θα πρέπει να γίνει σε επαφή με τους καταναλωτές και τον κλάδο της βιομηχανίας, τον κλάδο του τουρισμού, διότι έχουν αναπτύξει τα δικά τους συστήματα, τους δικούς τους καταλόγους που ήδη έχουν καρπούς στην αναγνώριση των ε, τίτλων ε, συμφωνώ απόλυτα. Αναφέρεται στο κείμενο. Ο κύριος Στεγκάντες ε, έχει υποβάλει συγκεκριμένες τοπολογίε σχετικά με την συνεργασία ανάμεσα σε διάφορες περιφέρειες, το ίδιο και ο κύριος Δανέλης και άλλοι. Είναι μια βασική πτυχή και θα πρέπει να τονίσουμε συγκεκριμένες περιφέρειες και ε, την διαφοροποίηση των τουριστικών προορισμών. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία αλλά και ανταγωνισμός ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες. Στο θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου και της διαβίου μάθησης συμφωνούμε ότι υπάρχουν πολύ καλές τροπολογίες σε αυτά τα θέματα και υπήρχαν και καλές τροπολογίες προηγουμένως στο θέμα των ε, διασυνδέσεων με διάφορες ε, περιφέρειες και νησιά. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, Πρόεδρε, ότι ο κ. Χάμερ και εγώ θα καταφέρουμε να βρούμε τη σωστή διατύπωση, το σωστό κείμενο κατά τη διάρκεια των μας διακοπών θα πρέπει να προσπαθούμε να μιλήσουμε για τον τουρισμό και την αηφορία. Θα πρέπει να βρούμε συμβαστικές τροπολογίες σε αυτά τα θέματα και ένα τελικό σημείο σε αυτά που είπε η κυρία Φώστερ για το σύστημα Καλύψο, τη δράση Καλύψο. Ε, πρόσωπος της Κομισιόν σας έδωσε την απάντηση νομίζω. Λυπάμαι αν άφησα κάτι πίσω, αλλά θα έρθω σε επαφή με τα αντίστοιχα άτομα τις επόμενες μέρες για περαιτέρω διευκρινήσεις. Οι τροπολογίες ήταν όλες πολύ θετικέ και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Φιντάντσα. Να υπενθυμίσω τα μέλη ότι η ψηφοφορία προβλέπεται ε, στην Επιτροπή ε, Μεταφορών Μαΐου και στις 2 Ιουνίου στην Ολομέλεια. έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινή μας μερίσιας διάταξης. Θα κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα και μετά θα κάνουμε συνάντηση των συντονιστών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη που τήρησαν τους χρόνους, διότι είχαμε τρία μεγάλα θέματα προς συζήτηση και καταφέραμε να κρατήσουμε τους χρόνους μας. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία.